Uh, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια ειδική συνάντηση αυτή μόνο για σήμερα. Έχουμε διάφορα σημαντικά θέματα και όλος ιδιαίτερος θέλω να καλωσορίσω εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα μας παρουσιάσει το επόμενο θέμα για την άθεση βάσεων παραχώρησης και σε κάποιο άλλο θα παρέμβει επίσης αργότερα. Έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πρώτα. Πρώτα απ' όλα ε, μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου, στο διαδίκτυο δηλαδή η συνεδρίασή μας, οπότε καλωσορίζω και οποιοδήποτε μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Ε, θα έχουμε και κάποιες παρουσίες που θα μπορέσετε να τις δείτε αργότερα. Στο μεταξύ ελέγχουμε και την ε, εμπειρία των ανθρώπων που μας παρακολουθούν κάθε στο διαδίκτυο. Οπότε πόσο, εφόσον θέλετε τις εμπειρίες σας να μας τις μεταφέρετε, στείλτε μας ένα mail. Ανακοινώσεις λοιπόν. Είχαμε συνάντηση, συγκρότηση σε σώμα, ήταν στις 23 Ιανουαρίου για την επανεκλογή μου. Στις 24 είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση μεταξύ των συντονιστών για να ασχοληθούμε με την μελλοντική μας οργάνωση τα επόμενα δυόμιση χρόνια, με το πρόγραμμα εργασιών μας, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό ε, νομοθετικό ε, πρόγραμμα μπροστά μας, το γνωρίζετε. Έχουμε... Σας έχουμε δώσει επίσης και ένα έντυπο που αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να οργανώνουμε τις συνεδριάσεις μας και τις εργασίες μας στο μέλλον, είναι και στο, στην ιστοσελίδα μας και υπάρχει και ένα άλλο έγγραφο πάλι στην ιστοσελίδα για τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Θέλω να καλωσορίσω τον αντιπρόεδρό μας, τον Τζίνο Τραματέρα, καλώς ήρθατε εδώ, ο οποίος δεν ήταν ε, την ε, ημέρα που είχαμε την συνεδρίαση συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής μας. Μήπως ε, θέλετε να πείτε δύο λόγια. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύντομα παίρνω το λόγο για να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη την οποία μου δείξατε ορίζοντας με αντιπρόεδρο στην ψηφοφορία της 25ης Ιανουαρίου στην οποία δεν μπόρεσα να πάρω μέρος όπως το είπε και ο πρόεδρος γιατί είχα προβλήματα υγείας. Πάντως σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να προχωρήσω με την ευθύνη την οποία που εναποθέσατε με κάθε δυνατότητα που έχω και με κάθε ικανότητα ελπίζω θα προχωρήσω. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ αλλά δεν ήταν από μένα εγώ το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Τρεματέρα. Ελπίζω να προχωρήσουμε σε μια καλή συνεργασία. Οι αντιπρόεδροι παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν θα έπρεπε να μην πω εδώ ότι πρέπει να ευχαριστήσω και την Προκάτω σα, την Λόρα Κόμη, η οποία ήταν, η Λάουρα η οποία ήταν αντιπρόεδρος και δυόμιση χρόνια και η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και αυτή πάντα. Ένας νέος Ιταλός αντιπρόεδρος λοιπόν θα συνεχίσει την καλή δουλειά. To Σχετικά τώρα με τις πρόορες δυνατότητες εξέτασης των θεμάτων με το Συμβούλιο. Ξέρετε ε, τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσαμε μέχρι τώρα και τις οποίες έχουμε επισημοποιήσει μέσω της αλλαγής ε, του κανονισμού. Εμείς δίνουμε πάρα πολλές δυνατότητες στον εισηγητή μας και τους σκιώδης με το Συμβούλιο, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εγκρίνει η εντολή φυσικά, την, να εγκρίνει η Επιτροπή τη συγκεκριμένη εντολή και το περιεχόμενο του, τε, του τεχνικής αν θέλετε λεπτομέρειας. Έχουμε δύο εκθέσεις που αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα, τα τρίκυκλα και τετράκυκλα όπως επίσης και τις ρυθμίσεις για γεωργικούς ελκυστήρες. Λοιπόν, η διαδικασία, η γραπτή που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα δείχνει ότι με μία εξαίρεση δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις συμφωνίες αυτές. Αυτό το οποίο απαιτείται όμως στα πλαίσια των νέων κανονισμών είναι να ψηφίσουμε τις συγκεκριμένες εντολές και άνω του 50% των μελών πρέπει να τις εγκρίνουν. Σας προτείνω λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχουν εκ νέου αντιρρήσεις, μετά τις ψηφοφορίες να βάλουμε το θέμα αυτό σε ψηφοφορία και να δώσουμε τη δυνατότητα στους εισηγητές ε, να επιβεβαιώσουν ή να πούν ότι άλλο θέλουν σε σχέση με την επιβεβαίωση της δικής τους εντολής. Ένα τελευταίο σημείο από τον Πρόεδρο. Ε, να πω ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ζήτησε από όλες τις επιτροπές να επανεξετάσουν τα χρονοδιαγράμματά τους γιατί θέλουν να προχωρήσουν σε μείωση του κόστους της διερμηνίας. Ε, οργανώνοντας συνεδριάσεις ε, δύο ομάδες επιτροπών ε, και τη Δευτέρα και την Πέμπτη και όχι μόνο την Τρίτη και την Τετάρτη. Ο υπεύθυνο των επιτροπών ασχολείται με τα θέματα αυτά και θα μας κάνει προτάσεις λόγω ακριβώς της πάρα πολλή δουλειά η οποία μας περιμένει, οι αλλαγές που προβλέπονται μειώνουν κατά τέσσερις συνεδριάσεις τις συνεδριάσεις μας σε αιτήσια βάση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν εμείς πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και να δούμε τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα πάντως να ζητήσω από όλους και από τους πολιτικούς συντονιστές να έχουν υπόψη τους ε, το θέμα αυτό. Έχουμε ορισμένες προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενία πράξη στα πλαίσια των οποίων υπό την Προεδρία του Βαν Ρόμποϊ το Συμβούλιο διευκρίνησε ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και είναι περίεργο, ε, μας ζητάνε να κάνουμε περισσότερα σε λιγότερο χρονικό διάστημα, το σημειώνουμε αυτό. Λοιπόν, θεωρώ ότι γίνεται δεκτή η πρόταση για την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν ε, κάποιες αλλαγές στους φακέλους σας. Υπάρχουν κάποια πρακτικά μάλλον, τα οποία θα θεωρηθούν δεκτά μέχρι το τέλος συνεδρίασης αν δεν υπάρξει κάποια εκπεφρασμένη αντίρρηση. Λοιπόν, ένα από τα θέματα αυτά είναι η τρίτη οδηγία σε σχέση με το τοπίο θα έλεγα των δημοσίων προμηθειών και αναθέσεων συμβάσεων παραχώρησης. Ο Φιλίπ Ζουβά είναι ο εισηγητής μας και θα ζητήσω και από τους κοιόδης εισηγητές αμέσως μετά να πάρουν το λόγο. Πρώτα όμως θα ακούσουμε την παρουσίαση την οποία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Τζοάννα Σικόρσκα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο θέμα αυτό. Θα μας κάνει και αυτή μια μικρή παρουσίαση και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους Σκιώδης και τον εισηγητή μας. Λοιπόν, αυτό είναι. Κύριε Ζούβα, θέλετε να κάνετε κάποια προκαταρκτική παρατήρηση ή να ζητήσει από την Επιτροπή να ξεκινήσει. Έχουμε εκπροσώπους του Συμβουλίου, βλέπω εδώ κάποιους γνωστούς από το Συμβούλιο εδώ, συμμετέχοντες και γι' αυτό θα περάσουμε αμέσως στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Σεκόρσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την πρόταση αυτή. Θα προσπαθήσω καταρχήν να σας εξηγήσω για ποιους λόγους προτείνεται το κείμενο αυτό. Και επίσης θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και την αρχιτεκτονική της πρότασης αυτής. Ξεκινάω λέγοντας ότι ο κύριος στόχος των ε, κανόνων όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Τέτοιο ίδιο ακριβώ ισχύει και εδώ, γιατί οι παραχωρήσεις επίσης επίπτουν στο ίδιο πλαίσιο. Υπάρχουν όμως διαφορές. Όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, μιλάμε για εξυγχρονισμό, για πιο αποτελεσματικούς κανόνες, ενώ όταν μιλάμε για παραχώρηση, τότε προσπαθούμε να θέσουμε τους βασικούς κανόνες ή με άλλα λόγια να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα στον ανταγωνισμό είναι τα ίδια όπως ισχύει και με τις δημόσιες συμβάσεις. Όταν λοιπόν κοιτάμε πώς έχει η κατάσταση στο παράγωγο δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, νομίζω ότι οι διαφορές φαίνονται. Οι δημόσιες συμβάσεις, εάν ε, ακούν στον κανόνα πώς γίνεται δημοσίευση, πώς γίνεται ανάθεση και πώς ε, ε, γίνονται διορθώσεις, τότε στην περίπτωση που έχουμε παραχωρήσεις για τις υπηρεσίες, δεν έχουμε παρά μερικώς μόνο ορισμένα πράγματα για κάποιου τομεί για τι υπηρεσίε δεν έχουμε τίποτα για παράδειγμα. Για τι ε, για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια. δεν έχουμε τίποτα απολύτω. ή δεν έχουμε παράγω δίκαιο καθόλου. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε το παραγωγό αυτό δίκαιο. Πρώτα απ' όλα για να διασφαλίσουμε ότι δαπανώνται καλά τα χρήματα, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων μπορεί να υπάρχει καλή πρόσβαση στις αγορές και επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι τέτοιοι κανόνες διευκολύνουν και την εταιρική σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, άρα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία βελτιώνουν με τη σειρά τους τις επενδύσεις και την καινοτομία. Επίσης, αξίζει τον κόπο να αναρωτηθούμε περί τίνος δεν πρόκειται όμως. Τι είναι αυτό που λείπει από την πρόταση. Και αυτό δείχνει γιατί αιτιολογείται και η πρόταση αυτή. Δεν πρόκειται μόνο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Αυτοί οι κανόνες δεν έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων σε κάποιον τομέα. Δεν θέλουμε σώνει και καλά οι δημόσιες υπηρεσίες να εξωτερικεύσουν την ανάθεση. Δεν πρόκειται δηλαδή για την αφισβήτηση της ποιότητας. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε οικονομικές δραστηριότητε. Είναι κανόνες που ισχύουν, θα ισχύουν στο μέλλον και δεν ισχύουν επί του παρόντος. Πριν καταλήξουμε σε πρόταση, προηγουμένως, προχωρήσαμε σε διάφορες μελέτες και προβαρασκευαστική δουλειά. Και νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο σημαντικές ε, διαδικασίες που ακολουθήσαμε πριν καταλήξουμε. Είχαμε δηλαδή μελέτες που πέρασαν και από τη δημόσια διαβούλευση. Πάνω από 60 διμερώς συναντήσεις έγιναν σε όλες τις χώρες ε, μέλη με όλους τους ενδιαφερόμενους. Με άλλα λόγια δηλαδή σε βάθος έγινε ανάλυση και των νομικών ε, στοιχείων και της γενικής κατάστασης. Εδώ βλέπετε κάποια νούμερα. Όχι όλα, κάποια από τόσες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγηση. 41% όσων απάντησαν λένε ότι υπάρχει πρόβλημα για την είσοδο στις αγοράς. Ε, σχεδόν 40% λένε ότι ξέρουν ότι, παρα... ότι η ανάθεση μάλλον γίνεται πολλές φορές ε, χωρίς να υπάρχει διαφάνεια 32% ε, λένε ότι υπάρχουν εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και 61,6% όσων απάντησαν λένε ότι η δημοσίευση των ε, κοινοποίησεων για παραχώρηση στην ε, επίσημη εφημερίδα θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια. Εδώ έχω να κάνω ένα επίσης σχόλιο. Οι εκθέσεις αξιολόγησης ήταν δύσκολες για έναν βασικό λόγο επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια, όπως σας είπα πριν, δεν υπάρχουν συστηματικά στοιχεία, συσσωρευμένα. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η αξιολόγηση αυτή είναι περιορισμένης ποιότητας και γι' αυτό και θέλαμε ευρεία διαβούλευση, γιατί θέλουμε με τους κανόνες αυτούς ακριβώς να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της έλλειψης της διαφάνειας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την αγορά και τις παραχωρήσεις. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να διακρίνουμε διαφόρων ειδών στρεβλώσεις. Έλλειψη ε, νομικής βεβαιότητας όσον αφορά τον ορισμό δηλαδή και την ανάθεση των ε, παραχωρήσεων, ε, την ύπαρξη εμποδίων κατά την είσοδο στην αγορά, είτε υπάρχουν πολύ διαφορετικοί κανόνες, είτε δεν είναι αρκετά συγκεκριμένοι, είτε γιατί οι πρακτικές των δημοσίων αρχών είναι διαφορετικές μεταξύ τους άλλοι είναι πολύ ε, σκληροί στην αντιμετώπιση τους, άλλοι όχι. Και τέλος δεν υπάρχει επαρκής νομική ασφάλεια, δικονομική εγγύηση δηλαδή, που σημαίνει ότι οι προσφέροντες δεν έχουν πάντα αρκετές εγγύσεις στην διάθεσή τους. Μερικές φορές δεν υπάρχει καθόλου ε, τέτοια εγγύηση. Είναι επίσης σημαντικό πιστεύω να σχολιάσουμε εδώ λίγο και τη σύμπτωση στα ευρήματα της μελέτης αυτής και της μελέτης που έγινε από το τμήμα πολιτικής του 2010 όπου το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών κατέληξε στο ίδιο ακριβώ συμπέρασμα, ότι το ότι δεν υπάρχουν κανόνες έχει σαν αποτέλεσμα οι νομοθεσίες στα κράτη-μέλη να είναι διαφορετικές και άρα να εφαρμόζονται διαφορετικές προδιαγραφές τέλος ότι ούτε οι οικονομικοί φορείς ούτε οι δημόσιες αρχές επωφελούνται από μια τέτοια κατάσταση διαφοροποίησης. Εμείς ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι έχουμε καταλήξει τα ίδια συμπεράσματα. Τι προβλέπετε λοιπόν. Τρεις ε, εναλλακτικές λύσεις. Βασικούς κανόνες, λεπτομερείς κανόνες και μικτούς κανόνες. Οι βασικοί κανόνες είναι αυτοί που εφαρμόζονται και σήμερα, οι οποίοι προσφέρουν κάποια διαφάνεια, αλλά δεν υπάρχει επαρκής δικονομική εγγύηση. Έπειτα υπάρχουν οι λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να, να απαντήσουμε στα σχόλια που λένε ότι οι σημερινοί κανόνες ε, δεν είναι ε, δεν είναι λεπτομερής όπως ε, πριν. Έπειτα υπάρχει και η τρίτη περίπτωση των μεικτών κανόνων που είναι ο καλύτερος συμβιβασμός ανάμεσα σε αυτά που υπάρχουν ε, σήμερα και στις παραχωρήσεις και στις δημόσιες συμβάσεις. Εδώ έχουμε κάποιες διατάξεις που έχουν να κάνουν με τους βασικούς κανόνες για την διαφάνεια. Έχουμε εγγυήσεις όσον αφορά τη διαδικασία, και προβλέπονται επίσης και τροποποίησεις. Κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι κι αλλιώς η αγορά το ήθελε αυτό. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην περίπτωση αυτή των παραχωρήσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτοί που θα υποφεληθούν είναι από τη μια μεριά οι αναθέτουσες αρχές και οι αρμόδιες αρχές με 82% των όσων απάντησαν να το επιβεβαιώνουν αυτόν. Στη συνέχεια είναι οι χρήστες που θα υποφεληθούν, επειδή θα είναι πιο χαμηλές ε, οι τιμές στην ίδια και τέλος οι επιχειρήσεις, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι η πρόσβασή τους στην αγορά θα είναι πιο εύκολη για τις παραχωρήσεις και αυτό το απάντησαν 83% των ερωτηθέντων. Έρχομαι τώρα στην αρχιτεκτονική της πρότασης. Ποια είναι η προσήκησή μας. Θεωρούμε ότι το πιο εύκολο θα ήταν να έχουμε έναν ενιαίο, ένα ενιαίο πακέτο κανόνων για τις παραχωρήσεις ότι είναι πιο εύκολο για τους χρήστες κάτι τέτοιο, αλλά και για τις συμβαλόμενες αρχές να έχουν ένα πακέτο κανόνων και γι' αυτό και αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό και για την κοινή ωφέλεια. Αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για την διευκόλυνση, πώς θα συγχωνεύσουμε δύο κείμενα. Εδώ πέρα μας ενδιαφέρει να αφαιρέσουμε και κάποιους κανόνες οι οποίοι δυσκολεύουν την ε, κατάσταση. Γιατί ακριβώς θέλουμε την απλοποίηση. Από την άλλη μεριά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο άρθρο είδαμε τι αποφάσει έχει πάρει και το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όσον αφορά τη διαφάνεια, για παράδειγμα, και στη συνέχεια τι αποφάσισε, τι, που έχει καταλήξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει της νομολογίας του. Το δικαστήριο μας βοηθάει να διατηρούμε τη συνοχή. Τέλος, ελαστικότητα. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, αλλά για μας ελαστικότητα σημαίνει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για τις ε, αναθέτουσες αρχές. Τι θα καλύπτει τώρα το μέτρο αυτό. Πρώτα απ' όλα όλες οι συμβάσεις παραχώρησης, 5 εκατομμύρια περίπου, θα ακολουθούν σε διάφορους κανόνες. Εδώ εξετάσαμε διάφορες περιπτώσεις σε διάφορους τομείς. 5 εκατομμύρια αποφασίσαμε και για τα έργα και για τις υπηρεσίες και για την κοινή ωφέλεια. Πρόκειται δηλαδή για παντός είδους παραχωρήσεις. Δεν καλύπτονται μόνο οι συνεργασίες δημοσίου-δημοσίου, ούτε περιλαμβάνονται τομεί οι οποίοι ήδη ρυθμίζονται από άλλου τομεακού κανόνε, μεταφορέ για παράδειγμα ή ενέργειε μεταφορέ. Και έχουμε και ειδικό καθεστώ για τι κοινωνικέ υπηρεσίε, ακριβώ επειδή υπακούν σε ειδικά χαρακτηριστικά. Μόνο η διαφάνεια ισχύει. Εδώ θέλω να σας εξηγήσω κάπως σύντομα για τον ορισμό. Έχουμε έναν ορισμό που σήμερα δεν είναι αρκετά σαφή. Το δικαστήριο το έχει πει πολλές φορές ότι δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο ενώ ο ορισμός που έχουμε τώρα είναι πια και εξηγούμε περί τίνος πρόκειται. Επίσης κάναμε και μία διευκρίνηση για να είναι ξεκάθαρο ότι οι άδειε δεν καλύπτονται από την οδηγία αυτή. Μιλάμε μόνο δηλαδή για συμβάσεις και όχι για άδειες. επιλέξαμε βασικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με ε, δημοσιεύσεις ex post και ex ante. Επίσης αποφασίσαμε να καθορίσουμε και τη διάρκεια των ε, παραχωρήσεων, χωρίς όμως κάτι συγκεκριμένο, επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία βάσο και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε για μία άδεια που να καλύπτει όλες τις παραχωρήσεις. Οπότε εξαρτάται και από τις επενδύσεις που γίνονται. Τέλος, επειδή ακριβώς ακούμε τι λέει η αγορά, θεωρήσαμε ότι οι κανόνες τροποποίησης ήταν κάτι αναγκαίο. Να υπάρχουν δηλαδή προβλέψεις για το πώς μπορεί ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο σύμβασης παραχώρησης να τροποποιηθεί. Δεν έχουμε ε, εγγύσεις διαδικασιών, είναι πολύ βασικό. Η οδηγία αυτή δεν περιλαμβάνει καμία διαδικασία. Οι μόνες εγγύησεις διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι προσφέροντες είναι ότι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν κάποια κριτήρια αποκλεισμού που εφαρμόζονται εύκολα και υπάρχει βέβαια και διάταξη για επανόρθωση εφόσον διαπιστωθεί κάποια στρέβλωση. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι ότι Σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς για τις παραχωρήσεις, ευελιξίες δηλαδή λοιπά, Έχουμε κάποια γενικά κριτήρια για την ανάθεση. Επιτρέπουμε επίσης και την εμπειρία και άλλα στοιχεία του προσφέροντος να ληφθούν υπόψη. Αυτό είναι κάτι καινούριο και που προσφέρει επιπλέον ευελιξία στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Τι σημαίνει τώρα μια πιο ελαστική προσέγγιση. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν υποχρεωτικές διαδικασίες, ότι δεν υπάρχουν ε, κανόνες ε, για τους ε, αναθέτοντας, δεν υπάρχουν ποσοστώσεις για υπεργολαβία και δεν υπάρχουν κανόνες που υπάρχουν σήμερα για τις δημόσιες συμβάσεις. Ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις. Τέλος για την ευελιξία υπάρχει και στα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού και ανάθεσης. Μιλήσαμε για την διάρκεια, ε, πέντε χρόνια αντί για δύο χρόνια που είναι για τις δημόσιες συμβάσεις και πιο ελαφριές διαδικασίες. Η πρόταση λοιπόν αντιμετωπίζει και δίνει λύσει σε προβλήματα που είχαν να κάνουν με την μη επαρκή πρόσβαση στην αγορά εξαιτία τη έλλειψη δικονομικών εγγύσεων. είναι κάτι που εφαρμόζεται εφόσον οι δημόσιες αρχές αποφασίζουν να αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε τρίτη πλευρά. Δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν δηλαδή, μόνο εφόσον το επιθυμούν. Τι πρέπει να κάνει τότε η αρχή υπαρχώς, να δημοσιεύσει μια κοινοποίηση, να ακολουθήσει κάποιους ε, κανόνες και τέλος, βάσει τη ρύθμιση αυτής, όλοι οι προσφέροντες μπαίνουν επίσης όρις. Δεν έχουμε διαφορετικές διαδικασίες δηλαδή. Τέλος, πιστεύουμε πως η οδηγία αυτή έχει την δυνατότητα να βοηθήσει και στην εξοικονόμηση δημοσίου χρήματο. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στο Συμβούλιο στις 17 Ιανουαρίου της ε, πρότασης αυτής. Με θετικές αντιδράσεις. Πολλοί ξεκάθαρα είπαν ότι είναι υπέρ και πολλοί άλλοι είπαν ότι είναι υπέρ του στόχου που καλύπτει η οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σαφέστατη είναι η παρουσίασή σας. Έχουμε βεβαίως και στην ιστοσελίδα μας την παρουσίασή σας, την έχουμε και εμείς. Και τώρα βεβαίως ο εισηγητής μας, ο κύριος Ζουβά, έχει το λόγο, η Σκιώδης, ο κύριος Αντσέρη από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες, η κυρία Ρούιλε, κύριος Διόν δεν είναι εδώ, Κόσιουσνετ, Σαμπίνη και Σφάμπ. Α, και ο κύριος Ταραμπέλα είναι παρόν. Εισηγητής για την άλλη οδικία για τις α, δημόσιες συμβάσεις, η κυρία Γκέπχατ επίσης και όποιος άλλος βεβαίως θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Ίσως έχουμε και χρόνο για κάποιες ερωτήσεις και στο τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Ζιβά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι για λόγους που ίσως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κατανοήσω, ενδεχομένως στο τέλος της συζήτησης να μπορέσω, διαπιστώνω ότι πρόκειται για ένα κείμενο που έχει προκαλέσει φόβο σε πολλούς. Κάποιοι δεν θέλουν καθόλου αυτό το κείμενο, άλλοι λένε ότι είναι απαραίτητο το κείμενο αυτό για την καλή λειτουργία αυτή της αγοράς. Άλλοι φοβούνται επιχειρήματα που δεν ε, περιέχονται στο κείμενο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πραγματικά ότι χρειαζόμαστε συζήτηση έτσι ώστε να διαλευκανθούν όλα αυτά τα σημεία. Πρώτη ερώτηση που θα έκανα είναι ποια είναι η χρησιμότητα αυτού του κειμένου. Και θα απαντούσα ότι πρόκειται για ένα κείμενο χρήσιμο, καθότι χρειαζόμαστε κοινού κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις συμβάσεις παραχωρήσεων. Μου φαίνεται λογικό. Όλοι θεωρούν, και ο κ. Ταραμπέλα και εγώ, και όλοι όσοι εργάστηκαν στο κείμενο αυτό, όλοι μας θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες και για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά και για τις συμβάσεις παραχωρήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κατηγορία εταιρικών σχέσεων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή δεν ιδιωτικοποιείται, αλλά παραχωρείται, ανατίθεται μία συγκεκριμένη υπηρεσία έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο δημόσιος τομέας. Αυτή η ανάθεση, αυτή η παραχώρηση γίνεται με χρηματοδότηση εν μέρη ή και χωρίς χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι η ανάληψη του κινδύνου τελικά γίνεται με ισορροπημένο τρόπο. Πρόκειται για μια μεταφορά κάποιων στοιχείων ευθύνης. Και θα πρέπει σαφώς να γίνει διάκριση εδώ μεταξύ των δημόσιων συμβάσεων και των ε, συμβάσεων παραχωρήσεων. Αλλά, ακόμα και αν δεν γίνει τόσο σαφή αυτή η διάκριση, όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειάζονται κοινοί κανόνες και για τις δύο αυτές περιπτώσεις και για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και για τις συμβάσεις παραχωρήσεων. Πολλές φορές επίσης βλέπουμε, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, ότι η δημιουργία υποδομών είναι κάτι που μπορεί να στηριχτεί σε εταιρικέ σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αν κάποιος από εμά ήταν δήμαρχος μιας κοινότητας, ενός δήμου, και θέλει να χρηματοδοτήσει μια δαπανηρή υποδομή με ένα χώρο στάθμευσης, παραδείγματο χάρη, αν η κοινότητα, ο Δήμος δεν έχει τους πόρους για να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει και το ρίσκο της εκμετάλλευσης. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το νομικό εργαλείο που να επιτρέπει αυτή την συνεργασία, αυτή την εταιρική σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει ε, βάσει κοινών κανόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να λειτουργήσουν με κοινούς κανόνες. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος ε, ιδιωτικός φορέας να πρέπει να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ε, απαιτήσει και να λειτουργήσει με διαφορετικούς κανόνες εάν βρίσκεται στην Ιταλία, στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός όσον αφορά την ομοθεσία και τελικά περιμένουμε την εξέλιξη της νομολογίας για να υπάρξει μία κοινή αντιμετώπιση. Είναι παράλογο αυτό. Κάθε φορά που ένας δήμος, ένας δήμαρχος, ένας επιχειρηματίας συνάπτει μία συμφωνία για ένα έργο, έχει τον φόβο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, ότι οι κανόνες θα αλλάξουν. Υπάρχει μεγάλη νομική αβεβαιότητα. Και θα δείξω και ένα άλλο σημείο. Πιστεύω ότι όσο προχωράμε στη συζήτηση τόσο θα καταλαβαίνουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Το άρθρο 26 παραδείγματος χάρη μου φαίνεται περίπλοκο. Χρειάζεται πρώτα μία γνωμοδότηση πριν την παραχώρηση, μετά πέραμε στην παραχώρηση, κατόπιν στην ανάθεση. Χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι περίπλοκο ακόμα το σύστημα. Παρόλα αυτά θα έλεγα ότι θα ήταν ακόμα χειρότερο να μην είχαμε τίποτα και να αφήναμε τα κράτη-μέλη να αναθέτουν πολύ σημαντικά έργα πολλές φορές βάσει ενός κανόνα αναπερίπτωση, όπως θα έλεγα, και άλλα κράτη τα οποία έχουν μια εξαιρετικά λεπτομεριακή νομοθεσία. Σκοπός μας συνάδελφοι, δεν είναι να ψηφίσουμε σήμερα εδώ μια επιπλέον οδηγία, αλλά να κάνουμε ένα βήμα προς ένα σύστημα ενιαίο, προς περισσότερη ομοιογένεια, προς ένα καινούριο κόσμο. Το ερώτημα είναι, προτιμάμε να αφήσουμε τον καθένα να συνεχίζει να κάνει όπως ξέρει, να μαγειρεύει στη γωνίτσα του με τον τρόπο που μέχρι τώρα έκανε και να ανατίθενται τα έργα με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, έχω βεβαίως πολλές ερωτήσει στην παρουσίαση της ε, Επιτροπής και γι' αυτό και θα σας πρότεινα, επειδή έχω πολλές ερωτήσει να υποβάλω ένα έγγραφο. Πείτε μου ποιε είναι οι προθεσμίε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Το θέμα όμως είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι θα προτιμήσετε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν θα αφήνει πολλά περιθώρια. Πρόκειται όμως για κάτι που σήμερα δεν το αντιμετωπίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστούμε χρόνο, πιστεύω. Ίσως δεν πρέπει να βιαστούμε αυτή τη φορά, γιατί πρέπει να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο, κοινά αποδεκτό κείμενο. Σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία για το κείμενο αυτό. Δώστε μας λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες. Από την άλλη μεριά βεβαίως καταλαβαίνω ότι θα πρέπει το χρονοδιάγραμμά μας να είναι παράλληλο με αυτό των δημόσιων συμβάσεων, γιατί πολλά θέματα συμπίπτουν. Ο ορισμός της παραχώρησης, παραδείγματος χάρη. Η παραχώρηση είναι κάτι που ουσιαστικά διακρίνει άλλου είδους συμβάσεις, διακρίνεται από άλλους είδους συμβάσεις, είναι το ρίσκο. Είναι το ρίσκο. Αυτό είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό, αν θέλετε, των παραχωρήσεων. Είναι κάτι, ένα στοιχείο νομικό, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μία κειμενόμενη, θα έλεγα, νομολογία. Το ρίσκο είναι ένα καθοριστικό στοιχείο, πώς μπορούμε να το ορίσουμε. Η Επιτροπή ομιλεί στο κείμενό της για ουσιαστική σημασία αυτού του χαρακτηριστικού, το ρίσκο. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για ιστορικούς λόγους και επειδή έχουμε ειδικέ περιπτώσεις ανάλογα με τις χώρες, ανάλογα με τις εθνικές νομοθεσίες, ανάλογα με τις τιμές που επιβάλλονται στη μία ή την άλλη χώρα, θα πρέπει να δούμε πώς θα οδηγηθούμε σε κάποια κοινά στοιχεία. Αυτό το 80-90% που βρίσκεται στην πρόταση, στο κείμενο, όσον αφορά την δημόσια δραστηριότητα. Αυτό μου φαίνεται μια λογική πρόταση. Επίσης, όσον αφορά το έργο, οι μεγάλες επενδύσεις, καθώς και ο χρόνος της παραχώρησης σε σχέση με κάποιες άλλες χρηματοδοτήσεις επιπλέον θα έλεγα. Και εδώ θα πρέπει να ξαναυπολογιστεί ο χρόνος παραχώρησης με ποιο τρόπο, με ποιους κανόνες. Όσον αφορά τις παραχωρήσεις ε, βάσει μιας ε, προηγούμενης, προηγούμενης συμφωνίας και αυτή η περίπτωση κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να συζητηθεί και να διαλευκανθεί. Πρόεδρος, ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα πρόταση. Έχουμε την σύμβαση για τις δημόσιες συμβάσεις και βεβαίως θα πρέπει να δούμε αυτή τη νέα πρόταση σε σχέση με αυτήν για τις δημόσιες συμβάσεις. Τώρα, οι σκιώδες. Σύντομα βεβαίως γιατί θα πρέπει να έχουμε τελειώσει στις 4. Ο κύριος Παντσάρη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πλήρως και γι' αυτό θα σταματήσω μόνο σε συγκεκριμένα από τα θέματα που έχουμε εδώ. Καταρχάς στο ερώτημα το οποίο δεν έθεσε ελπίζω θεωρητικά ο κ. Ζουβέν η νομολογία αυτή είναι επίκαιρη για μια σειρά θα έλεγα από αιτίες τις οποίες ελπίζω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν και κάποια άλλα θυμία στα οποία η πρόταση αυτή οδηγίας νομίζω πρέπει να αναλυθεί περισσότερο. Υπάρχει ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στην οδηγία αυτή και στην οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε πολύ και το οποίο για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία σχετικά με τις κοινωνικές ρήτρες. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι αν από τη μία ζητάμε περισσότερους διακανονισμούς και ρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό, δεν είναι σαφές πώς η οδηγία αυτή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Σαν παράδειγμα την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, το θέμα της συλλογή των απορριμμάτων και επίσης, διαρωτώ με αν έχει λάβει υπόψη η μελέτη επιπτώσεων τις κοινωνικές επιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχουν αναφορές στην ποιότητα της εργασίας, στο δικαίωμα διαβούλευσης, στη σύνοψη συλλογικών συμβάσεων και τη συμμετοχή γενικότερα των εργαζομένων στη διαδικασία. Ο κύριος Μπαρνιέ σας θυμίζω ότι είχε πει ότι αυτά τα θέματα δεν θα τα αγνοήσει. Υπάρχει επίσης και το θέμα του ορισμού του κινδύνου και αυτό είναι κεντρικό θέμα σε σχέση με τη διάκριση ανάμεσα σε σύμβαση παραχώρησης και σε δημόσια προμήθεια ή δημόσια σύμβαση. Το 2.2 το νομίζω δεν δίνει την απάντηση την κανονική σε σχέση με τον κίνδυνο ο οποίος αναφέρεται εκεί. Η απάντηση δεν είναι σαφής, είναι επιφανειακή και πρέπει να διευκρινιστεί ακόμα περισσότερο. Και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, σύμπτωσης σε κάποιους τομείς της εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας με την οδηγία για τις προμήθειες. Υπάρχουν ερωτηματικά λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε και ακόμα περισσότερα. Πού σαν παράδειγμα θα μπορέσουμε να ταξινομήσουμε ορισμένε από τις υπηρεσίες. Σαν παράδειγμα τις ε, παραχωρήσεις άδεια λειτουργίας ε, θερινών ε, καταλημάτων ή λουτρών κτλ. Εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι το πολύ επιλεκτικό χαρακτηριστικό της δυνατότητας που έχουν τα κράτη-μέλη να επιλέγουν ε, την συγκεκριμένη ή όχι διαδικασία είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει με να επιτρέψουμε στις δημόσιες διοικήσεις να ακολουθήσουν διαδικασίες πιο ευέλικτες αλλά να μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένες μορφές ε, νομικής ρύθμισης. Θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις επίσης, ε, εγγυήσεις για τη διαφάνεια στους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να ελέγχουν τις διαδικασίες αυτές. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοήσει η Επιτροπή. Και υπάρχει και το θέμα της διάρκειας. Η διάρκεια μιας παραχώρησης καθορίζεται με πολύ γενικό τρόπο. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι λόγος ε, θα έλεγα διάκρισης ε, εις βάρος του ενός ή του άλλου επιχειρηματικού παίκτη. Και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν μελέτες επιπτώσεων σε σχέση με τις πιθανές επιλογές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο χρήζει επίσης εμβάθυνσης είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο νομίζω για όλους. Είμαστε όλοι διαθέσιμοι όμως. Ευχαριστώ κύριε Παντσαρή. Ο κύριος Μάντελς θέλει να πάρει το λόγο από τους ε, φιλελευθέρους. Όχι, η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να στον κύριο Ζουβά όταν έθεσε το ερώτημα γιατί χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο εκθέσεις αυτής της Επιτροπής. Οι ρυθμίσεις που προσπαθούμε εδώ να υιοθετήσουμε έχουν άμεση σχέση με τις τρευλώσεις ε, του ανταγωνισμού στην αγορά και τα αποτελέσματα και ε, ερωτηματολογίων αλλά και ερευνών που έχουν γίνει δείχνουν ότι σήμερα δεν είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε με ακρίβεια. Μας λείπουν στοιχεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε αν όντως υπάρχει στρέβλωση σε αυτό το τομέα ναι ή όχι. Δεύτερον, υπάρχει μια εμπειρία 40 χρόνια τέτοιων παραχωρήσεων και συμβάσεων και οι έρευνες που έχουν γίνει όταν αναφερόμαστε στην ασφάλεια του δικαίου, στην ε, νομική βεβαιότητα κτλ, θα πρέπει πραγματικά να βασιστούμε στα πραγματικά στοιχεία αυτού του παρελθόντος, αυτών των 40 ετών, για να δούμε ακριβώς τι ακριβώς πρέπει να γίνει σε σχέση με τις ε, ρυθμίσεις και τους κανονισμούς που υιοθετούμε για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις δημόσιες παραχωρήσεις όσον αφορά τον τομέα των παραχωρήσεων, των συμβάσεων παραχωρήσεων. Δεν είναι σαφή τα πράγματα και επίσης δεν είναι σαφής οι ορισμοί όλων αυτών των ενιών. Αυτό για μένα είναι καθοριστικό. Ας βασιστούμε λοιπόν στο παρελθόν, στην εμπειρία του παρελθόν, για να δούμε πώς θα στηρίξουμε και, τους δύο αυτούς, και τις δύο αυτές προσπάθειες ρύθμισης. Ο κύριος Ζουβά αναφέρθηκε στον ρόλο του δημόσιου τομέα και αναρωτιέμαι γιατί στις δημόσιες συμβάσεις ιδιαίτερα στην πολύ σημαντική ακρόαση που οργανώσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα και σε απαντήσεις για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά με λυπεί ιδιαίτερα και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να το ε, κάνει. Όσον αφορά την αρχή της ε, αναλογικότητας, δηλαδή του τι είδους ε, ρύθμιση και κανονισμούς χρειαζόμαστε, αν θα πρέπει να η Επιτροπή παίρνει μια παράξενη θέση για το θέμα αυτό και αναρωτιέμαι. Πώς ελήφθη υπόψη εδώ η αρχή της αναλογικότητας. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτός ο κανονισμός εδώ ξεπερνάει τι αρμοδιότητες και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει τέτοιου είδους ρύθμιση. Ιδιαίτερα θεωρώ ότι δεν απλοποιείται η διαδικασία για την σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί η εταιρική σχέση μεταξύ παραδείγματος χάρη ενός Δήμου και ενός ιδιωτικού φορέα και θα συνεχίσει η ρύθμιση όπως γίνεται μέχρι τώρα. Πρόεδρος. Ο κύριος Διό, βλέπω ήρθε. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Βεβαίω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομο θα είμαι. Ζητώ συγγνώμη καταρχήν, διότι καθυστέρησα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα από αυτό που μόλις άκουσα. Γιατί θυμάμαι συζητήσεις που είχαμε προηγουμένως για το ίδιο θέμα σε αυτήν την Επιτροπή και πολλοί βουλευτές εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, έλεγαν ότι πραγματικά δεν χρειαζόμαστε καμία πρόταση κανονισμού, γιατί διότι μας αρκεί η νομολογία του δικαστηρίου. Τελικά υπάρχει πρόταση, υπάρχει πρόταση Επιτροπής και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον εγώ θα συνεισφέρω, είμαι καταρχήν από αυτούς που θέλουν να διαπιστωθεί η ανάγκη μιας τέτοιας ε, νομοθεσίας. Ε, και αφού πιστώ γι' αυτό, αφού πιστούμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, τότε να προχωρήσουμε σε αρχές όπως η αναλογικότητα, η επικουρικότητα, που βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε σε ποιο επίπεδο θα δράσουμε. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα. Βλέπουμε βεβαίως ότι η Επιτροπή έχει εργαστεί, ότι έχει προχωρήσει η πρόταση της Επιτροπής. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει στις χώρες μας να εξηγήσουμε ότι χρειάζονται επιπλέον κανονισμοί γιατί η Επιτροπή θέλει περισσότερη διαφάνεια. Και αυτό, όπως ξέρετε, δεν θα είναι εύκολο να το εξηγήσουμε. Πρόεδρος. Προς το παρόν εγώ δεν θα σχολιάσω, ίσως στο τέλος της συζήτησης θα δούμε. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές, παρακαλώ πάρα πολύ σύντομοι. Και μετά θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει απαντήσεις. Γιατί μιλάμε για την εισαγωγική συζήτηση νομίζω ότι επί τη βάση του κειμένου εργασίας του κ. Ζουβά θα επανέλθουμε σε λεποπτέρειες. Βάιλαντ. Κυρία Βάιλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, έχω τρεις ερωτήσεις. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι μια πρώτη γενική συζήτηση. Θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα που είναι οι πολιτικοί σε τοπικό επίπεδο θα μπουν στην ουσία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ενσωματώνονται εδώ βεβαίως και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ενώ ακούσαμε ότι δεν εμπεριέχονται στο κείμενο της ε, οδηγίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε οι κοινωνικές υπηρεσίες εδώ πώς ορίζονται. Θα θέλαμε να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί εμείς βεβαίως δεν θέλουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες στην ε, οδηγία. Δεύτερη ερώτηση. Δεν ανυψώσατε το όριο για τις υπηρεσίες στη συζήτηση που είχαμε τις προηγούμενες φορές, τις δύο προηγούμενες εκθέσεις και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα των 5 εκατομμυρίων λέγοντας ότι είναι πολύ χαμηλό το όριο και ότι θα θέλαμε να είναι πιο υψηλό το ανώτατο όριο για για τις υπηρεσίες. Γιατί λοιπόν παραμείνατε σε αυτό το σχετικά χαμηλό ποσό των 5 εκατομμυρίων. Τρίτη ερώτηση, κάτι που επίσης με ξάφνιασε πολύ, το ζητήσαμε και διμερός. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι υπηρεσίες στα λιμάνια θα έπρεπε να αποκλειστούν. Ξέρετε την κατάσταση στα λιμάνια, όχι μόνο στη Γερμανία, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν αποκλίνονται αυτές οι υπηρεσίες. Ο κύριος Φάμπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στον εισηγητή όσον αφορά το σχολιασμό για την μελέτη αντικτύπου. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα σχόλια, αλλά θα ήθελα εγώ προσωπικά να επανέλθω στο θέμα. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία πραγματικά δεν είναι μια πρόταση που γίνεται κοινά αποδεκτή. Και η ερώτηση γιατί αυτή η πρόταση είναι χρήσιμη δεν είναι σαφής. Εγώ προσωπικά θα απαντούσα ότι πολλά σχόλια άκουσα και είδα, πολλά ερωτηματολόγια, πολλές δημοσκοπήσεις, αλλά αυτά δεν αρκούν, δεν είναι επαρκής βάση για να προχωρήσουμε σε αυτή την πρόταση. Δεύτερον, αυτά τα 5 εκατομμύρια, κάνετε την ερώτηση όσον αφορά το όριο, Έχω την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει η δημόσια υποχρέωση για τις ε, συμβάσεις αυτών των 5 εκατομμυρίων. Το ποσό αυτό δηλαδή υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο οι εταίροι μας φυσικά και θα μας επικρίνουν εάν αλλάξουμε αυτό το ποσό. Και νομίζω ότι ακριβώς για αυτό το λόγο βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική δυσκολία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να αυξηθεί αυτό το όριο και να μην παραμείνει στο όριο που ισχύει για όλες τις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις. Αλλά πραγματικά επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα, υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζουβά για την εισαγωγή, την παρουσίαση που μας κάνατε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, κάνατε μια πολύ σωστή παρατήρηση με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι για αυτού του είδους τα θέματα χρειαζόμαστε χρόνο. Υπάρχουν δυσκολίες, είναι περίπλοκο το θέμα και πρέπει να ε, το συζητήσουμε έτσι ώστε να ρυθμιστούν σοβαρά ερωτήματα. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με αυτό που είπατε, ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και όσο και να θέλουμε να βιαστούμε, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι για αυτό το θέμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο χρόνο. Δεύτερον, η ομάδα μου έχει πει και στο παρελθόν για το θέμα αυτό των παραχωρήσεων ότι θα πρέπει να βασιστούμε στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Εάν δηλαδή το δικαστήριο είχε πάρει κάποιες τέτοιες αποφάσεις, να βασιζόμασταν σε αυτά. Τίποτα τέτοιο όμως κατά την απόψή μου δεν έχει γίνει και ουσιαστικά εμείς εδώ θα συζητήσουμε πάνω σε μια ανύπαρκτη βάση. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα των παραχωρήσεων όχι μόνο σε θέματα κοινωνικών υπηρεσιών αλλά γενικότερα σε θέματα υπηρεσιών κοινή ωφελία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ μας λέει η Επιτροπή ότι δεν συμπεριλαμβάνονται. Υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις ε, που αποκλείουν. Το ερώτημα όμως είναι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Εάν υπάρχουν πρέπει να ξέρετε ότι η δική μου πολιτική ομάδα θα έχει πάρα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις και δυσκολίες. Θα θέλαμε πραγματικά να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι διάβασα προσεκτικά το κείμενο το βρίσκω πάρα πολύ περίπλοκο. Δεν μου φαίνεται ότι δεν είναι γραφειοκρατικό και είναι και ασαφές. Και όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας του δικαίου, δεν νομίζω ότι πετυχαίνουμε κάτι παραπάνω με το κείμενο αυτό. Διαβάζοντάς το, δεν κατάλαβα πραγματικά για ποιους Τομεί υπηρεσιών, για ποιες κατηγορίες υπηρεσιών ισχύει και για ποιους όχι. Και αν δεν ξεκαθαρίσουμε αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία του κειμένου. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να κάνουμε αυτό. Και κάνω την ίδια ερώτηση με την κυρία Βάιλερ εδώ. Σε συζητήσεις που είχαμε με τον Επίτροπο Μπαρνιέ, είχα την εντύπωση ότι οι υπηρεσίες ε, που αφορούν τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι σε μια διαφορετική κατηγορία. Από το κείμενο δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω ότι αποκλείονται. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να επεξεργαστούμε το κείμενο. Αν θέλουμε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη βεβαιότητα δικαίου, θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ, να αλλάξουμε το κείμενο αυτό και να ρυθμίσουμε μόνο τους τομείς που χρήζουν ρύθμισης. Και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε οι, υπηρεσίες κοινωνικής, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας να είναι μέσα ε, στην ε, οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε διαφορετικά θέματα από εκείνα τα οποία συζητούσαμε στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που υπήρχαν αλλαγές, μάλλον που εδώ υπάρχουν αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα οδηγία. Έχει δίκιο πάντως ο εισηγητής που λέει ότι χρειάζεται να δούμε πού υπάρχουν θεμελιώδες ε, αλλαγές. Η κυρία Σικόφσκα, σας απαντήσει, παρακαλώ. Θα την προσκαλέσουμε φαντάζομαι και κάποια άλλη στιγμή για να ξανασυστήσουμε, αλλά και τώρα αν μπορεί ας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις τόσο σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλες. Θα αρκεστώ στα πιο σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα γιατί χρειαζόμαστε αυτούς τους κανόνες. Επανέρχομαι στο πρώτο το οποίο σας ε, είπα, που ήταν ότι η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης αποτελεί μέρος των ε, δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή είναι ένας τρόπος που δαπανούνται ε, που το δημόσιο χρήμα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να έχουμε υπόψη μας και την ίση μεταχείριση μεταξύ όλων εκείνων που υποβάλλουν προσφορές. Ένα πράγμα θα προσθέσω σε αυτό. Αν δούμε πώς ε, μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τις ε, δημόσιες συμβάσεις, ένα από τα στοιχεία ήταν να καταργήσουμε τους κανόνες. Αλλά καταλήξαμε στο ότι θα ήταν πολύ χειρότερο αυτό και από πλευρά διαφάνεια και από πλευρά αφήνεια και από πλευρά πρόσβαση στι αγορέ και θα υπήρχε ένα πλήρε νομικό κοινό. Γι' αυτό θέλουμε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα στι ε, παραχωρήσει. Τώρα για τα πιο συγκεκριμένα ερωτήματά σα. Κομισιόν οργάνωσε δύο ευρείες διαβουλεύσεις και με επιχειρήσεις και ατομικά με Το καλοκαίρι του 2011 για παράδειγμα έγινε ε, μελέτη επιπτώσεων η οποία βασίστηκε σε ευρεία διαβούλευση με την κοινή γνώμη. Για το κείμενο το πόσο είναι περίπλοκο ή όχι. Οι κανόνες είναι περίπλοκοι γιατί η ε, συμβάσεις είναι ένα περίπλοκο θέμα. Προσπαθούμε όμως να απλοποιήσουμε χρησιμοποιώντας μόνο τους κανόνες εκείνους οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι αναγκαίοι. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα εδώ τα πράγματα από ότι με τις δημόσιες συμβάσεις. Αν υπάρχει κάποιο πεδίο βελτίωσης, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, δεν Για το κατά πόσο καλύπτονται κοινωνικές υπηρεσίες ή όχι. Σήμερα οι κοινωνικές υπηρεσίες καλύπτονται από το παράρτημα Β και ειδικού κανόνες, όπως για τις δημόσιες συμβάσεις. Εδώ πήγαμε ένα βήμα πιο πέρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται από κανένα διαδικαστικό κανόνα της ε, οδηγίας αυτής, μόνο υπάρχει υποχρέωση για εξάντε και εξ post ενημέρωση. Είναι το μόνο όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές. Για τις κοινοφιλείς υπηρεσίες τώρα η οδηγία δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις οικονομικού τύπου ή άλλες. Μιλάει για όλες τις υπηρεσίες αυτές στην αγορά. Για τους λιμένες τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα στις υπηρεσίες ε, λιμένος. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που συνδέονται με την παραγωγικότητα. Κάποιες θα καλύπτονται, κάποιες δεν θα καλύπτονται. Και γιατί, γιατί αυτό θα εξαρτάται από το γενικότερο σκηνικό. Δεν καλύπτονται όλες ε, λοιπόν οι υπηρεσίες στη γη, για παράδειγμα. πρέπει να έχετε υπόψη σας, δηλαδή ότι οι υπηρεσίες στους λιμένες θα καλύπτονται ε, κατά περίπτωση. Δεν μπορούμε να πούμε γενικά ναι ή όχι. Εξαρτάται από τη νομική μορφή. Για τα όρια τώρα, τα κατόφλια, τα εξετάσαμε με διάφορες τιμές και καταλήξαμε στο ότι για έργα και υπηρεσίες βάσει συμβάσεων ε, ανατομέα, έχοντας κοιτάξει τις διάφορες περιπτώσεις, θεωρήσαμε ότι τα 5 εκατομμύρια είναι το σωστό επίπεδο. η παραχώρηση υπηρεσιών δεν καλύπτονται από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το στοιχείο δηλαδή. Α, ναι. Ένα τελευταίο για την ομολογία. Μπορεί να είναι εκτενής αλλά όχι πλήρης. Οπότε αν ρωτήσετε τι είναι η παραχώρηση, πώς δημοσιεύεται και πώς ανατίθεται, θα πάρετε 27 διαφορετικές απαντήσεις όσες και οι μέλη. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε, να έχουμε έναν ορισμό και μία δέσμη υποχρεώσεων όσον αφορά τις παραχωρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μας βοηθήσατε με την παρουσίασή σας. Σίγουρα θα μας δοθεί και πάλι ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αναφέρατε την μελέτη που ανέθεσε η δικιά μας επιτροπή, ήταν έργο της κυρίας Ρούλε. Δεν ξέρω, ελπίζω να το έχουν πάρει όλοι οι βουλευτές. Κύριε Ζουδά, θα ξαναβρεθούμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας πάλι και περιμένω το έγγραφο εργασία σας. Οπότε κλείνουμε εδώ το θέμα, και αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι βέβαια. Ναι, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πρώτον, αντίθετα με τις εντυπώσεις που δείχνουν ότι είμαστε πολύ μακριά εμένα από τους δε, αυτό δεν ισχύει, γιατί συμφωνούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και την ομολογία, αλλά και να την ελέγχουμε αυτήν, γιατί μερικές φορές υπάρχουν αντιφάσεις. Και εγώ πολύ θα ήθελα να υπάρχει ένα κείμενο κωδικοποίησης της νομολογίας, αλλά δεν γίνεται γιατί υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στην ομολογία. Για τις υπηρεσίες συμφωνώ και εγώ με την ερώτηση της κυρίας Γκέπερτ, πρέπει να το δούμε. Τέλος. Αν στόχος είναι να υπάρχει και απλοποίηση και νομική ασφάλεια, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και νομίζω, Πρόεδρε, ότι δείξαμε όλοι ότι χρειάζεται ακόμα χρόνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνεισέφεραν στη συζήτηση αυτή. Έχουμε τώρα μια άλλη σημαντική νομοθετική πρόταση. Πρόκειται για την τελωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοτική ιδιοκτησία. Εισηγητή είναι ο κύριο Γιούργεν Κρότσμαν. Η κυρία Καρολάιν Έντερη επίση είναι εδώ, που είναι επικεφαλή ε, του τμήματο για την ε, θέση σε εφαρμογή των μέτρων αυτών. Στόχος μας σήμερα το απόγευμα είναι να ακούσουμε τον κύριο Κρότσμαν για τις 199 ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στο σχέδιο έκθεσης. Είχαμε τροπολογίες μάλιστα και από άλλες επιτροπές, όπου όμως εμείς βάσει του άρθρου 50 έχουμε την αποκλειστική αρμοδιότητα. Σίγουρα θα αναφερθείτε και σε αυτές τις τροπολογίες. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ πέρα συντάκτες νομοδοτήσεων. Όχι. Ωραία. Ο κύριος Κρότσμαν πρώτα θα πάρει το λόγο, μετά οι σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Γκάλο, η κυρία Χέντ είναι εδώ. Ο κύριος Έγκστρομ σίγουρα, η κυρία Μακλάκεν και ο κύριος Δε Θα κάνουμε το γύρο αυτόν, αλλά προηγουμένως ο εισηγητής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ. Στην ε, έκθεσή μου Υπήρξαν αρχικά 71 τροπολογίες. Θα κάνουμε και εδώ την προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ μας. Εννοείται ότι υπάρχουν και μερικά επίμαχα ζητήματα, δεν το αρνούμε αυτό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μερικά από αυτά. Και εγώ υπέβαλα τροπολογίες υπό το φως των συζητήσεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας προκειμένου να βοηθήσω στην εξέβρεση ενός συμβιβασμού. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για τις παράλληλες ε, παράνομες εισαγωγές. Εδώ προσπάθησα να πετύχω κάποια συμφωνία. Εμένω στη θέση μου πιστεύω ότι κάθε παραβίαση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να καταδικάζεται ακόμα και οι παράλληλες εισαγωγέ. ανεξάρτητα από ποιο δίκιο κοιτάμε, το εθνικό ή όχι. Οι παράλληλες εισαγωγές είναι παράνομες, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για σήματα για τα οποία υπάρχει σε εθνικό επίπεδο προστασία ακόμα και αν δεν έχουν μπει στην αγορά άλλων χωρών τα προϊόντα αυτά, επειδή δεν έχει υπάρξει ακόμα άδεια για αυτά. Ορισμένοι λένε πως όχι, εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Είναι επιπλέον δουλειά για τα τελωνία και ε, περιορίζει και όλα τον... την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο αποτελεσματικό στα σύνορα να σταματάμε τα προϊόντα παρά να περιμένουμε να κυκλοφορήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, οι αρχές, όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον κίνδυνο κάθε φορά που ελέγχουν προϊόντα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής. Τα προϊόντα έτσι κι αλλιώς ελέγχονται. Και όσοι λένε ναι, αλλά δεν ευνοεί αυτό τον καταναλωτή, εγώ λέω με προσοχή, γιατί οι παράλληλε αγωγέ δεν είναι ίδια ποιότητα όπω και τα αυθεντικά προϊόντα, άρα μπορεί να τεθεί πρόβλημα δημόσια υγεία και σύγχυση στο μυαλό του καταναλωτή. Υπέβαλα λοιπόν εγώ τροπολογίες με τις οποίες συμπληρώνω την πρότασή μου σε κάποια σημεία και έλαβα υπόψη μου μάλιστα και τις αντιδράσεις που είχα μέχρι τώρα πιο συγκεκριμένα για τις τροπολογίες. Στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, εγώ εξήγησα για ποιο λόγο πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να ακούμε τους εισαγωγείς. Άλλοι είπαν, ε, μα όχι εδώ είναι θέμα απόφασης δικαστηρίου. εκείνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι θίγονται ζωτικά του συμφέροντα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ακουστούν. Εγώ δεν πιστεύω όμω ότι η απόφαση αυτού του δικαστηρίου ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Έτσι κι αλλιώ εδώ πέρα μιλάμε για προσωρινά μέτρα που παίρνουν οι τελωνιακέ αρχέ μέχρι να έχουν επαληθεί ε, επαλυθεί τα γεγονότα πρέπει να έχουμε κάποιο περιθώριο χρονικό για να δούμε κατά πόσο παραβιάζονται τα δικαιώματα δυνατικής ιδιοκτησία ή όχι. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια οριστική απόφαση όσον αφορά τι εισαγωγέ. Εννοείται ότι κάποια στιγμή στη διαδικασία θα έχει το δικαίωμα να ακουστεί ο ενδιαφερόμενο. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχουν 10 μέρε για ένσταση μετά από την ανακοίνωση της ε, απαγόρευσης ε, παρετέρω εισαγωγής του προϊόντος. Το άτομο δηλαδή μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης των τελωνιακών αρχών. Μην ξεχνάμε επίσης ότι οι τελωνιακές αρχές αντιδρούν πάντα κάθε φορά που υπάρχει υπόνοια, ε, με κάποια βάση βέβαια. Όταν δεν έχει κάνει ακόμα ένσταση, ο ενδιαφερόμενος. Συνήθως πρόκειται για την περίπτωση πειρατείας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αν υπάρχει μη βάσιμη υπόνοια από πλευράς των τελωνιακών αρχών. Το πρόβλημα τίθεται περισσότερο για τα διπλώματα βρεσιτεχνίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ψευδείς δηλώσεις δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση εξαιτίας του ανταγωνισμού για θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Και βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό είναι να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταχρηστικές διαδικασίες. Βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό είναι τα, να ρυθμίσουμε τις περιπτώσεις εμπορευμάτων τα οποία απλώς περνούν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προστατεύσουμε παραδείγματος χάρη τις ε, περιπτώσεις αυτών που κάποια μηχανήματα απλώς περνούν. Το θέμα δεν είναι να δούμε αν τα και τα προϊόντα Nokia και Philips απειλούνται από προϊόντα που έρχονται από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να δούμε πώς μπορεί με μια πολύ συγκεκριμένη υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις αυτών των εμπορευμάτων πάντα βασιζόμενοι στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Επίσης ε, υπάρχει και το θέμα της τροπολογίας που έχει υποβληθεί όσον αφορά την, ε, το βάρος Πρόκειται για περιπτώσεις ε, που δεν έχουμε αρκετές αποδείξεις, αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ότι πρόκειται για εμπορεύματα τα οποία ουσιαστικά θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ο τελικός ε, αποδέκτης είναι ένα κράτος τρίτο. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αυτές τις ε, περιπτώσεις εμπορευμάτων, όπως παραδείγματος χάρη τα γενώσιμα φάρμακα, τα οποία τελικά φαινόταν ότι απευθύνονται στη Λατινική Αμερική ήταν όμως τελικά εμπορεύματα τα οποία θα παρέμεναν σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα παράδειγμα τέτοιων καταχρήσεων. Αυτό που ιδιαίτερα μας απασχολεί εδώ είναι να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα εμπορεύματα και να αντιμετωπίσουμε παραδείγματο χάρη τις απομιμήσεις προϊόντων. Είναι αν θέλετε επίσης και το θέμα των ε, διαμεσολαβητών, των μεσαζόντων και εδώ τροποποίησα το αρχικό μου κείμενο όσον αφορά τις παραδείγματος άνοιες πεσμένες διαδικασίες για τους ε, ενδιάμεσους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε τα άτομα αυτά ή τις εταιρείες ή τους φορείς Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεταφορεί είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται και πρέπει να κάνουμε κάποιου μαύρους καταλόγους, μαύρες λίστες. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια τροποποίηση. Έχω βάλει και κάποια νέα στοιχεία βεβαίως στο κείμενο. Έλαβα υπόψη μου όλα αυτά που ακούσαμε, ιδιαίτερα για την προστασία των δεδομένων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων βεβαίω μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα και έχω βασιστεί και στις προτάσεις της Επιτροπής. Κοιτάξτε εδώ την τροπολογία μου. Η νομική βάση. Η νομική βάση έχω βασιστεί εδώ στην δημιουργία, στην ίδρυση μιας τράπεζας δεδομένων. Βεβαίως αυτό δεν υποστηρίζεται από την πρόταση της Επιτροπής. Και πιστεύω επίσης ότι οι τελωνιακές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται όταν υπάρξουν ε, κάποιες ε, υποψίες για καταχρήσεις και όταν δεν μπορεί η τελωνιακή αρχή να εντοπίσει τα άτομα, τις εταιρείες και σε αυτή την περίπτωση θα κρατούνται τα εμπορεύματα εάν μέσα στον απαραίτητο χρόνο που είναι 24 ώρες δεν μπορεί να εντοπιστεί ε, ο φορέας ε, ή το άτομο στον οποίο απευθύνονται τα εμπορεύματα. Για κάποιες επικίνδυνες ουσίες, για χημικές ουσίες, και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταχείες διαδικασίες για να μην καθυστερούν ε, τα εμπορεύματα, ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία βεβαίως σήμερα δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη και τα οποία θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν και να πολλαπλασιαστούν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα και να δημιουργηθούν ε, τράπεζες δεδομένων. Εδώ έχουμε θέσει και κάποιες προθεσμίες το 2013. Αυτά δεν έχω άλλες τροπολογίες. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες με θετικό πνεύμα για να φτάσουμε σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο. Επαναλαμβάνω, μείωση της γραφειοκρατίας για τις τελωνιακές αρχές και καλύτερη συνεργασία. Αυτές είναι οι δύο κατευθυντήριες ιδέες που θα ήθελα να ενισχύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρόιτσμαν. Οι εισηγητές, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις συμβαστικές τροπολογίες βεβαίως, θα σας κάνουν τις προτάσεις. Ξέχασα να σας πω ότι και η κυρία Γκάλο είναι ε, η εισηγήτρια εξ ονόματος της νομικής επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν υποβληθεί 259 τροπολογίες. Και εγώ όμως είμαι πολύ αισιόδοξη, όπως και ο εισηγητής, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Έχουμε προβλέψει και μία συνεδρίαση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών την το πρωί. Και πιστεύω ότι τα περισσότερα δύσκολα σημεία θα ξεπεραστούν. Συμβιβαστικές τροπολογίες θα υπάρξουν όσον αφορά την απλοποιημένη διαδικασία για τις απομιμήσεις, είναι το άρθρο 20, καθώς και η διαδικασία όσον αφορά τις παραβιάσεις ε, των ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησία, δηλαδή το άρθρο 23 και εδώ θα υπάρξει συμβαστική τροπολογία γιατί υπάρχει μια πρόταση του κυρίου Κρόιτσμαν που προτείνει η απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 για αυτές τις ε, περιπτώσεις απομιμήσεων να επιβληθεί σε όλες τις περιπτώσεις παραβιάσεων της νοηματικής ιδιοκτησίας. Θεωρώ επίσης ότι είναι απαραίτητος ο έλεγχος των εμπορευμάτων που περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό βεβαίως διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το νόμιμο εμπόριο δεν αφορά όλα αυτά τα προϊόντα και τις απομιμήσεις. Και θεωρώ βεβαίως ότι εδώ θα μας στηρίξει και η Επιτροπή. Όσον αφορά τα μικρά, τις μικρές αποστολές, πρόκειται για το 1383, εδώ απλοποιείται ακόμα περισσότερο η, η απλοποιημένη αυτή διαδικασία και πιστεύω ότι και εδώ θα υπάρξει συμφωνία. Τώρα, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες που μειώνουν λίγο την ε, ευθύνη, την ανάληψη ευθύνης από μέρους των ε, ενδιαμέσων και των μεταφορέων. Ένα σημείο για το οποίο δεν υπάρχει συμφωνία είναι οι παράλληλες εισαγωγές. Για το θέμα αυτό έχω πάρει το λόγο πολλές φορές στο παρελθόν. Και κάθε φορά που έχω πάρει το λόγο, υπενθύμησα ότι οι περισσότερες τελωνιακές αρχές των κρατών μελών είναι αντίθετες. Αυτό έχω διαπιστώσει. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Και αυτό βεβαίως για πολλούς λόγους. Γιατί οι τελωνιακές αρχές πρώτον θα αποκτήσουν επιπλέον ε, φόρτο εργασίας, θα πρέπει κάθε φορά να ελέγξουν τις συμβάσεις μεταξύ δύο επιχειρήσεων με δική τους ευθύνη. Και σήμερα οι τελωνιακές αρχές μας λένε ότι δεν είναι αρμόδιες και δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να επαληθεύσουν και να ελέγξουν όλες αυτές τις συμβάσεις. Δεν έχουν τις νομικές, αν θέλετε, τη νομική αρμοδιότητα. Αυτό που θέλουμε σήμερα είναι να υπάρχει μία αποτελεσματική και γρήγορη επέμβαση των τελωνιακών αρχών. Εάν λοιπόν δυσκολέψουμε περισσότερο και επιβαρύνουμε αυτές τις διαδικασίες, φτάνουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει παραβίαση μιας σύμβασης, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε εθνικό επίπεδο. Άρα η παρέμβαση των τελωνιακών αρχών δεν είναι απαραίτητη κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να μην συμπεριλάβουμε τις παράλληλες ε, εισαγωγές. Βεβαίως ο διάλογος θα συνεχιστεί ε, και θα υπάρξει και αυτή η συνάντηση που σας ε, προανέφερα των εισηγητών, των σχεδόν εισηγητών. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κατάλαβα ότι στη νομική επιτροπή έχετε ήδη ψηφίσει για την γνωμοδότησή σας. Ναι, στη Νομική Επιτροπή ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς. Κυρία Γκέπχαρτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Χέτ δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Ζητά συγγνώμη και μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω. Το κάνω ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω κάποια από τα σημεία που μου έχει επισημάνει. Έχει βεβαίως εμπλακεί προσωπικά και επίσης ζήτησε να αποκλειστούν από την οδηγία αυτή οι προσωπικές αποστολές γιατί πρόκειται για ένα θέμα που έχει ρυθμιστεί από άλλες οδηγίες. Τώρα, για τις παράλληλες εισαγωγές εδώ θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις ε, από μέρους ε, του εισηγητή ε, και του ΕΛΚ. Για πολλούς λόγους που δεν θέλω εδώ να επαναλάβω, θεωρώ ότι εδώ γίνεται πολύ πιο περίπλοκο το θέμα και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι τελωνιακές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να αναλάβουν αυτό το τομέα. Τώρα, για τα γενώσιμα φάρμακα. Θα πρέπει να ελέγξουμε, να υπάρχει ελεύθερη μεταφορά, ότι τα προϊόντα αυτά θα περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εμπόδια και όπως ξέρετε για τις απομιμήσεις, απομιμήσεις φαρμάκων υπάρχουν εδώ διάφορες τροπολογίες που ακούσαμε ότι θα τις υποστηρίξει και ο εισηγητής. Όσον αφορά την αντίστροφη του βάρους απόδειξης, συμφωνούμε με την πρόταση που υπάρχει στην τροπολογία. Συμφωνούμε επίσης με τον εισηγητή όσον αφορά τον ορισμό των λεγόμενων μικρών αποστολών. και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει αυτό να το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να υπάρξει ένας σαφής ορισμός που θα γίνει εκ των προτέρων από εμάς, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αβεβαιότητα. Και έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το θέμα αυτό ο εισηγητής. Η κυρία Χέντ θέλει επίσης ε, να υπογραμμίσει ότι το θέμα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να συζητηθεί. Όσον αφορά δηλαδή την ανάληψη κάποιου μέρους της ευθύνης. Όσον αφορά την απόδειξη, παραδείγματος χάρη για την προέλευση και την τελική αποστολή κάποιων εμπορευμάτων, τα αποδεκτικά στοιχεία, η ενδιάμεση, οι μεταφορείς και η κατανομή της ευθύνη Εδώ όλο αυτό το θέμα χρειάζεται περισσότερο συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ για τα σημεία που θέσατε. Έγκστρομ έχεις δει στο λόγο. Θα ήθελα να πω διάφορα, αλλά το βασικό είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην έκθεση αυτή έτσι ώστε να μην θα έλεγα αλωτριωθούμε από θέματα τα οποία μας είναι πολύ σημαντικά όπως η ελευθερία διακίνησης, η πίστη μας στα ελεύθερη αγορά κτλ. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα την κατάσταση μέσω επιμέρους ρυθμίσεων, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα για το νόμιμο εμπόριο. Έτσι και αλλιώς το παράνομο εμπόριο δεν θα τα λάβει αυτά υπόψη του. Οπότε όταν αλλάζει ο νόμος επηρεάζονται ελάχιστα αυτές οι παράνομες ενέργειες, περισσότερο επηρεάζονται οι νόμιμοι. Uh, I don't want Για τις προσωπικές αποσκευές έτσι και αλλιώ έχουν την δυνατότητα οι αρχές να ελέγχουν και ε, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το ε, τηλέφωνο το ασύρματο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια εγώ δεν θα ήθελα να δω να γίνεται και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξαιρέσουμε τις προσωπικές αποσκευές για τις μικρές αποστολές, πολλές μικρές αποστολές. Ξέρετε ότι οι καταναλωτές αγοράζουν κάτι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν δώσουμε τη δυνατότητα στα τελωνία να προχωρούν σε κατασχέσεις προϊόντων τυχαία λιγάκι, έτσι θα το βλέπαν οι καταναλωτές, τότε δημιουργούμε προβλήματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτή η τυχαία έλεγχη τι σημαίνει. Δεν είναι παράνομο για ένα καταναλωτή να εισάγει κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα σε διπλώματα επιστεχνίας γιατί το, οι νομικές συνέπειες ενός διπλώματος έβρεση τεχνίας δεν αφορούν τον καταναλωτή αλλά αφορούν τους εμπορικούς παίκτες, τους εταίρους. πάρα πολύ συχνά ο καταναλωτής πέφτει θύμα εγκληματικών δραστηριοτήτων και όχι δεν διαπράττει ο ίδιος κάποια τέτοια ενέργεια. Λοιπόν, θα πρέπει να δείξουμε σε σχέση με τις μικρές αποστολές ότι υπάρχει σωστή ενημέρωση ε, με τον σωστό τρόπο από το τελωνίο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, έτσι ώστε να γνωρίζει τουλάχιστον ο καταναλωτής περί τίνος πρόκειται και θα πρέπει να έχει και χρόνο έτσι ώστε να διαμαρτύρεται ή να ζητήσει να αποζημιωθεί ίσως. Το να περιμένει πάρα πολύ καιρό ε, δεν είναι επαρκές για τον καταναλωτή ο οποίος για πρώτη φορά θα πάρει ένα τόσο περίπλοκο γράμμα από τις αρχές του τελωνίου. Για τις παράλληλες εισαγωγές συμφωνώ με την κυρία είναι νόμιμες, πρέπει να είναι νόμιμες και όπως και να έχουν τα πράγματα δεν είναι αυτό το οποίο μας αφορά άμεσα. Εμείς μιλάμε για τον τελωνιακό κανονισμό και τις σχέσεις του με τα δικαιώματα τα πνευματικά, τα συγγενικά. Σχετικά την ευθύνη των ενδιαμέσων, σήμερα ποιες είναι οι βασικές αρχές. Όταν πραγματικά κάτι δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν δικαιούται κανείς να ελέγξει. Αυτό το κάνει για να προστατεύσει κάποια δικαιώματα τα οποία έχει, κάποιες προσω... κάποια προσωπικά δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα. Λοιπόν, οι αρχές ε, δεν είναι το θέμα να ρυθμίσουμε εμεί ότι δεν έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν κάποια πακέτα και δεν θα πρέπει εκεί που δεν είχαν την δυνατότητα αυτή εμείς να την εγκαταστήσουμε την έλλειψη αυτή με μια υποχρέωση να κάνουν τους ελέγχους. Δεν έχει λογική ε, σαν παράδειγμα για τις εταιρείε οι οποίες κάνουν τις μεταφορές. Δεν μπορούν να ελέγχουν οι εταιρείε αυτές ε, το περιεχόμενο των δεμάτων κτλ. Και εδώ είπαμε να μην φύγουμε τις νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες. αν είσαι μια εγκληματική οργάνωση και χρησιμοποιείς ενδιαμέσους για να φέρεις εις πέρας ε, τις, τις σκοπιμότητές σου, ε, αυτό είναι κάτι που δεν θα σε ενοχλήσει οι νέες ρυθμίσεις. Αυτοί οι οποίοι θα ανησυχήσουν είναι οι νόμιμοι εισαγωγή και μεταφορής. Ελπίζω λοιπόν να ανησυχήσετε κι εσείς όπως εγώ. Η κυρία Μακράκιν είναι η επόμενη. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή με τον οποίο εν πολύ συμφωνώ σχετικά με τον κώδικα για τα τελωνία κτλ. Ε, σύμφωνο ότι πρέπει να ενισχυθεί η έκθεση, θα συναντηθώ μαζί του, αλλά να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω, όπως λέω και στην πρώτη μου τροπολογία, απαιτείται καλύτερη συνεργασία και σωστή εφαρμογή ε, του τελωνιακού κώδικα. Και τα συστήματα τα τελωνιακά πρέπει να είναι διαλειτουργικά θα έλεγα για τον ορισμό για τις μικρές αποστολές, τα μικρά δέματα και τα λοιπά Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χάσουμε περισσότερο χρόνο, αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν θα πρέπει εμείς να επιβαρύνουμε επιπλέον <clears throat> τα δημοσιονομικά μιας χώρας σε σχέση με την λειτουργία των τελωνίων διότι και τα τελωνία θα πρέπει να χρησιμοποιούν επιπλέον προσωπικό για να κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους και να φέρνεις πέρα σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση παρανόμων δραστηριοτήτων. και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά σε σχέση με όλους όσους συμμετέχουν στη συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα η οποία παραβιάζει τους κανονισμούς. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο τελωνιακός κώδικας μερικές φορές δεν επιβάλλεται να εφαρμοστεί από τους ενδιαμέσους και τους μεταχωρείς. Έχω καταθέσει και άλλες τροπολογίες λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερες καθυστερήσεις απλά θα δώσουμε χρόνο ίσως για να καταστρέψουν παράνομα στοιχεία κάποιες εταιρείε, οι οποίες έχουν ασκούν παράνομες δραστηριότητες ελπίζω να έρθουμε σε επαφή για περισσότερες συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες θα προστατεύσουν τα συγγενικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για την ομάδα μου είναι σημαντικό η πρόταση αυτή να καταλήξει σε μια πρόταση η οποία θα βοηθήσει να υπάρξει και εξοικονόμηση πόρων. Εξού και οι τροπολογίες τις οποίες ε, υποβάλλουμε και εμείς σχετικά με τις προτερότητες για τους ε, ελέγχους οι οποίοι έτσι καλώς δεν μπορεί να γίνονται στο 100%. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα όπου βέβαια να βλέπουμε κατά πόσο έλεγχοι αξίζουν τον κόπο. Και μία από τις περιπτώσεις όπου τίθεται αυτό το δίλημα είναι για τις μικρές ή μεγάλες αποστολές. Τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία του καταναλωτή. μην ξεχνάμε ότι ο καταναλωτής πολλές φορές αγοράζει προϊόντα και μέσω του διαδικτύου. Αυτό το καταναλωτή δεν θα πρέπει να τον δυσκολεύουμε υπερβολικά με οχλήσεις. Και αυτό είναι μια κριτική που έχουμε εδώ. Για τις παράλληλες εισαγωγές αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. περισσότεροι όμως είπαν ε, ότι ήθελα να πω κι εγώ σχετικά με την οδηγία αυτή πρέπει να είναι εξαίρεση. Γιατί υπάρχουν τα γενώσιμα φάρμακα που δεν πρέπει να εμποδίζουμε την εισαγωγή τους. Έχω μια ερώτηση όμως στον κύριο Κράτσμαν για την άκτα. Ο τρόπος με τον οποίο θέλει άκτα να χειριζόμαστε τα γενώσιμα φάρμακα. Κύριε Κράτσμαν, Νομίζετε ότι υπάρχει συμβατό ανάμεσα στην πρόταση την εδώ και την άκτα. Right, I think we don't want to open a discussion on ACTA this afternoon, but our colleagues on Inter... Θα το κοιτάξει και ίντε σίγουρα. Και εσείς έχετε κάτι, παρακαλώ. Έχουν υποθεί αρκετά. Συμφωνήσω για την ανάγκη που υπάρχει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η πραγματική, θα έλεγα, η ουσιαστική εφαρμογή των προβλέψεων για να βοηθήσουμε και τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς, ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι πέφτουν θύματα παράδεκτων πρακτικών. Συμφωνώ λοιπόν να ορίσουμε σωστότερα τα προϊόντα πάνω στα οποία θα πρέπει να ασκούνται έλεγχοι γιατί φυσικά δεν έχουν όλα τα προϊόντα τον ίδιο θα έλεγα το ίδιο ποσοστό επικινδυνότητας κατά τα άλλα συμφωνώ σας ευχαριστώ λοιπόν νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η συζήτηση και των τροπολογιών Τώρα θα ακούσει και άκουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρότσμαν να κλείσει τη συζήτηση. Θα έχετε μία συνάντηση κύριε Κρότσμαν με τους σκιώδεις εισηγητές για να εξετάσετε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και ε, στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχουμε ε, γύρω από το άρθρο 50 και τις τροπολογίες των υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών γιατί ξέρετε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο πακέτο. Πάντως έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα σε όλους τους συναδέλφους να πω ότι παραδείγματος χάρη σαν την ευθύνη για τους ε, ενδιάμεσους το θέμα αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την υπάρχουσα τροπολογία. Τώρα, τα προσωπικά προσωπικές ε, αποσκευές. Το θέμα είναι ότι αυτό ρυθμίζεται από μία άλλη οδηγία και δεν θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και να το συζητήσουμε γιατί θα στείλουμε ένα λανθασμένο μήνυμα ουσιαστικά. Ο κόσμος δεν θα ξέρει ποια είναι η οδηγία που ρυθμίζει το θέμα αυτό. Τώρα για τις απομιμήσεις βεβαίως ε, όλοι είμαστε κατά και όλοι θέλουμε να περιοριστεί αυτή η δραστηριότητα. Δεν μιλάμε όμως ε, στο κείμενο αυτό για αυτές τις ε, περιπτώσεις μόνο. Η Επιτροπή και η Γερμανία θέλει να παραμείνει το, ο τομέας αυτό στην Επιτροπή. Το θέμα είναι εγώ τι έκανα. Προσπάθησα να υπερασπιστώ το κείμενο της Επιτροπής, διότι συμφωνώ τώρα. Αν δεν θέλει η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θέλουν οι σοσιαλιστές και δεν θέλει το ΕΛΚ, δεν θα μείνει αν μόνο η Γερμανική Επιτροπή. Το θέμα των γενώσιμων νομίζω έχει ρυθμιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εντοπίσουμε στο κείμενο. Όλοι συμφωνούν για τα γενώσιμα και βεβαίως ε, θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν χωρίς εμπόδια και χωρίς καθυστερήσεις τα φάρμακα αυτά εκτός Ευρώπης, στην Ινδία, στην Λατινική Αμερική και οπάνε. Τώρα, 28 Φεβρουαρίου ήταν η ημερομηνία και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Μάιο. Και συνάδελφοι, προσέξτε αυτές τις ημερομηνίες και πρέπει να πιέσουμε αν θέλουμε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και αν θέλουμε οι τελωνιακές αρχές να εργαστούν με λιγότερο γραφειοκρατικό άχθος, προσέξτε και το θέμα της επεξεργασίας των δεδομένων. Στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο περίπλοκα. Okay, well, thank you very much for that. Yes. Θα σε ευχαριστώ πολύ, με ο Πρόεδρος. 29 Φεβρουαρίου μάλλον θα ψηφίσουμε, έτσι μου λέει η γραμματεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει 28-29 στην ίδια εβδομάδα. Η κυρία Φερ, εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ξέρω ότι το θέμα προχωράει ικανοποιητικά. Ναι εντάξει. Ήθελα να πω ότι ήμουν στην ε, Κοπενχάγη την προηγούμενη εβδομάδα και άκουσα από μέρους ε, του Υπουργού ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ θετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήταν όλοι οι σκιώδεις παρόντες. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, συνεισφορές σας στη συζήτηση ψηφοφορία για την γνωμοδότηση της κυρίας Ιάνοβα. Είναι το επόμενο θέμα. Τρόφιμα για παιδιά, για βρέφη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικού ιατρικούς σκοπούς. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Βεβαίως, κυρία Ιβάνοβα, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Επίσης και οι σκιώδεις Εάν όμως κανείς δεν θέλει να πάρει το λόγο θα πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Κύριε Ιβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία και την ανταπόκρισή τους. Υπήρχαν αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία επέστησαν την προσοχή μας. Καταρχάς ο ορισμός διαιτητικού τροφίμου, τι ακριβώς σημαίνουν τα, τρόφιμα αυτά, τα τρόφιμα δυνατίσματος, δεν νομίζω ότι στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας να υπάρχει επαρκής νομική προστασία των καταναλωτών στα διάφορα κράτη-μέλη, όπου μέσω μιας απλής ανακοίνωσης ένα ή οδήποτε προϊόν μπορεί να αποκτά ένα τίτλο. Αυτό δεν δίδει επαρκή επίπεδα προστασίας του καταναλωτή. Μέσω της κατάργησης αυτών των ετικετών και για τα γάλατα για τη μικρή ηλικία κτλ. Υπάρχει βελτίωση της κατάστασης και θα απαιτηθούν πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις και συγκεκριμένες απαιτήσει για να υπάρξει τέτοιου είδους ε, χαρακτηρισμός του τροφίμου. και θα διατηρήσουμε το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και θα κρατήσουμε φυσικά ε, και θα βοηθήσουμε τη βιομηχανία. Νομίζω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σήμερα η Επιτροπή μας θα δείξει ότι υποστηρίζει αυτό το καλύτερο επίπεδο ε, προστασίας του καταναλωτή αποδεχόμενη όλες τις ομαδικές ψήφους και με τις ε, δίαιτες ε, χαμηλές θερμιδικά επίσης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Γραμματεία η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και επέδειξε ένα τεράστιο επαγγελματικό πνεύμα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, φυσικά θα συμφωνήσω και με την τελευταία σας παρατήρηση. Λοιπόν, οι σκιώδεις εισηγητές θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για τη συνεργασία την οποία επέδειξε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Υπάρχουν προφανώς δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές ε, θα φανούν ίσως σε κάποιες από τις ψήφους, αλλά στις περισσότερες συμφωνούμε. Η κυρία Παρβάνοβα. και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για την εξαιρετική της δουλειά. Η γνωμοδότηση αυτή θυμίζω ότι είχε γίνει αντικείμενο επεξεργασία σε επίπεδο τεχνικό στο παρελθόν μετά από διάφορες πιέσεις που δεχτήκαμε από τα λόμπι. Πάντα η προτεραιότητα την οποία δέχεται και η συγγήτρια είναι η προστασία του καταναλωτή όμως και είναι και απόλυτα συμβατή θα έλεγα με τις θέσεις και τη φιλοσοφία του κύριου ε, εισηγητή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ελπίζω να βελτιώσουμε την έκθεσή του. Ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα. Λοιπόν, κάποιος άλλος και όδης εισηγητής θέλει το λόγο. Όχι. Α, κύριος Σταβίνη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Τα πράγματα αλλάζουν σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν δεν κατάλαβα καλά και κάποια πράγματα, αλλά ε, η Ιταλική Ένωση ε, ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από ε, δυσανεξία στη γλουτένη είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από την κατάσταση αυτή γιατί πιστεύουν και δεν είναι δική μας γνώμη αυτή αλλά είναι δική τους γνώμη γιατί έχουν ειδικού που εργάζονται στον τομέα αυτό ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει σε κίνδυνο όλες ε, τις, όλα τα κατορθώματα θα έλεγα ε, τα οποία είχαν πετύχει οι ασθενείς αυτοί γιατί πρόκειται για ασθενείς δεν πρόκειται για επιλογές όπως η φυτοφάγη ας πούμε και πιστεύουν ότι η οδηγία αυτή θα λειτουργήσει εις βάρος τους και είναι διαμετρικά αντίθετη με τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό λοιπόν αποδεχόμενοι αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί στον τομέα βλέπω ότι από την ασθενεία αυτή της ανεξίας στην γλουτένη υποφέρουν 5 εκατομμύρια περίπου πολίτες. Quanto proposto, entrando nel merito uno per uno degli emendamenti ε, ελπίζω να δεχτούν την τροπολογία μας γιατί είναι μια τροπολογία η οποία είναι υποστηρίξιμη κυρίως και τεκμηριωμένη επιστημονικά και όχι τόσο πολιτικά. We Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα θα ήθελα να πω ότι ο κατάλογος που έχουμε μπροστά μας είναι διαφορετικός από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε ομαδικές ψήφους μετά από διαπραγμάτευση των εισηγητών και συνεισηγητών και σκιωδών εισηγητών μάλλον και βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει μετά από την κατάληψη της ψηφοφορίας κάθε φορά. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές ότι είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, η πρώτη ομαδική ψήφος, τρόφιμες εξειδικευμένης διατροφής. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος αμέσως. Άρχεται η ψηφοφορία η πρώτη ομαδική ψήφο στον κατάλογο που έχετε μπροστά σας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καλυφθούν από τη συγκεκριμένη αυτή πρόταση κανονισμού. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ομαδική ψήφο για ακριβώς ε, τους, ε, αυτούς που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Αν ψηφίσουμε υπέρ σημαίνει ότι ε, συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα αυτά. Άρχεται η ψηφοφορία για την δεύτερη αυτή κατηγορία προϊόντων τροφίμων. ...39 έχουν ψηφίσει... Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται και αυτή η πρόταση. Και τώρα περνάμε στην τρίτη ομαδική ψήφο για τα τρόφιμα με μειωμένη ενέργεια που προορίζονται για δίαιτες αδυνατίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία για τον κατάλογο ακριβώς αυτών των ε, τροπολογιών. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται συνολικά. Το 98 και 61 καταπίπτουν. Περνάμε τώρα στην ομαδική ψήφο για ορισμένα τρόφιμα αδυνατίσματος για το αν θα συμπεριληφθούν ή όχι στην πρόταση. Άρχεται η ψήφος. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε τώρα στην τροπολογία 68, 69 και 70 πιτέλα και σαλτίνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Για 68, 69 και 70. Τέλος. Απερίφθη περνάμε τώρα στα 71, 72 και 73 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτές. 74. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έχουμε άλλη μία ομαδική ψήφο για όλες τις τροπολογίες που ζητούν τη, τη συμπερίληψη ε, των γαλακτοκομικών που προορίζονται για νέα παιδιά. γάλακτος μάλλον για μικρές ηλικίε. Τέλος της φοφορίας, απερίφθη η πρόταση αυτή. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο μπλοκ τροπολογιών στην σελίδα 12. Ε, προϊόντα και τρόφιμα τα οποία ε, θα έλεγα οδηγούν σε αύξηση της μυϊκής μάζας εν Λοιπόν, Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Προχωρούμε στην τροπολογία 85, Βάισκεμπα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και μετά τροπολογία 11, Ιβάνοβα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε στην επόμενη ομαδική ψήφο, για δίαιτες με χαμηλά, ε, χαμηλές θερμίδες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Είναι δεκτές οι προτάσεις αυτές. Συνεχίζουμε με τις τροπολογίες 12 και 101. Ιβάνοβα και Παρβάνοβα. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτές. Έχουμε επίσης άλλη μια ομαδική ψήφο μετά σχετικά με τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και άλλες ουσίες που προστίθενται. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται, απορρίπτονται. Συνεχίζουμε με την 109 και 110. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτές. Η 13 τώρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά δεκτή. Η 14 ποιοι είναι υπέρ. Κατά δεκτή. Η 113 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οι 118 και 119 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτές. Η 120 σαν προσθήκη, ποιοι ή μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 120. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. 22 υπέρ, 18 κατά. Σαν προσθήκη. 122 και 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων. Τώρα ψηφίζουμε την 126 σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Η 122 τώρα, 123 και 124 ταυτόσημες ποιοι είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. Θέτουμε σε ψηφοφορία την 125 κατά διέρεση ψήφος εδώ. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτές. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα στην τροπολογία 16 Ιβάνοβα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 17 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα η 129 σε ψηφοφορία. Σαλβίνη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 135 και 137. Άρχεται η ψηφοφορία για το 135 και 137. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτονται. 136 τώρα Σαλβίνη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται 139 πιτέλα ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 18 τώρα ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή συμβιβαστική 3 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 141 Βερνιό ποιοι είναι υπέρ ή μάλλον ηλεκτρονική ψήφος για την 141 Βερνιό Πέρα στις ψηφοφορίες. Θα πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία γιατί δεν άφησα χρόνο για να ψηφίσουν όλοι. Λοιπόν, ψηφίζουμε εκ νέου την τροπολογία Βερνιό 141 ηλεκτρονική ψήφος. Νόμιζα ότι θα είχατε ψηφίσει περισσότεροι, έκανα λάθος. Πέντε δεν ψήφισαν. Λοιπόν, απορρίπτεται. 18 υπέρ, 22 κατά. 143 της εισηγήτριας, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. 151 και 152, ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 153 και 154, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Η 19 της εισηγήτριας, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 19 Πέραση ψηφοφορίας. Είναι δεκτή η 19. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ηλεκτρονική ψήφος για τη συμβιβαστική τροπολογία 2. πέρας της Νομίζω ότι δεν έχουν ψηφίσει ποτέ τόσοι πολλοί, 41 ψηφίσουν, 22 υπέρ, 19 κατά. Γίνεται δεκτή η συμβιβαστική 2. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική 3. Ή μάλλον του εισηγητή την 3, της εισηγήτριας την 3. Ξεκινάει η ψηφοφορία. δεκτή 28 υπέρ 13 κατά 36 Παρφάνοβα ποιοι είναι υπέρ για μια στιγμή λέει α, ο πρόεδρος άλλα λέει ο κύριος Βάμπα αλλά κάνω τα μέλη του 36 λέει τώρα ο πρόεδρος 36 είναι υπέρ κατά δεκτή Οπότε καταπίπτει το άλλο κείμενο. Τροπολογία 4 της ηγήτριας. Υπέρ, κατά, δεκτή. 43 και 45. Ψηφίζουμε την 43 και 45. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτονται. 6 της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 50 τώρα. Προσθήκη. Προφορική τροπολογία. Δεκτή γενικά. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Καταπίπτει η κανονική 50. 48 και 49. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Η 55 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τοπολογία 7 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. πέρασε της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τώρα η 63 κοράτσα μπίλτ. Είναι, υπάρχει μια προφορική τροπολογία εδώ θα την καταθέσει κάποιος είναι μάλλον κάποιος κατά της κατάθεσης αυτής όχι, η συγγήτρια. Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι και σε σχέση με τις υπόλοιπες τροπολογίες λέμε ότι για να διορθωθεί η κατάσταση το γάλα που προορίζεται για παιδική τροφή θα πρέπει να ενταχθεί στην 194 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ισχυρισμούς που πρέπει να περιλαμβάνονται στα τρόφιμα τα οποία κυκλοφορούν. σύμφωνα με τον κανονισμό 1169 του 2011 του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2009 1925 του 2006 και της αποφάσεως της 20 Σεπτεμβρίου του 2006 για την προσθήκη ίχνων και μετάλλων στα τρόφιμα και της Οδηγίας 2046 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και της αποφάσεως της 10ης Ιουνίου για την σύγκληση των νομικών ρυθμίσεων των κρατών μελών. Λοιπόν, είχατε καμιά αντίρρηση για αυτά που ακούστηκαν. Εντάξει λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για αυτήν την προφορική τροπολογία. δεκτή 26 υπέρ 15 κατά. Καλό θα ήταν για όλα αυτά να κάνει κανείς ε, υποσημειώσεις και όχι να τα συμπεριλαμβάνει στο κείμενο με προφορική τροπολογία. Λοιπόν, η 10 της εισηγήτριας, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. 65 και 66, ποιοι είναι υπέρ, κατά απορρίπτονται 67 της εισηγήτριας ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτές περνάμε τώρα στην τελική ψήφο άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Ο 41ος θέλει να ψηφίσει και αυτός. Όχι. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας. 35 υπέρ και μία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα. Θα υπερασπιστείτε σωστά τη θέση μας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ και τα 41 μέλη που ήταν εδώ και λάμπριναν με την παρουσία του στη συνεδρίασή μας. Περνάμε τώρα στην τροπολογία της κυρίας Κόρχολα. So I äh, Κύριε Πρόεδρε, είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής η κυρία Κόρολα, αλλά βρίσκεται στην Φιλανδία, πρέπει να παραστεί σε μια σημαντική επέτειο και γι' αυτό και σήμερα δεν θα μπορέσει να είναι εδώ. Αλλά πιστεύω θα βρεθούν ε, λύσεις ε, για τα ακόμα επίμαχα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ισκιώδης, δεν θέλει κανείς το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε με τις τροπολογίες. Πρόκειται για την περιαγωγή στα δημόσια δίκτυα. Ξεκινάμε με την 95 τροπολογία. Ξεκινάμε. Τροπολογία 95. Τέλος. Απορρίπτεται. 96 της Χέτ. Αρχή της ψηφοφορίας. 96. Τέλος. Απορρίπτεται επίσης. 98, ταραμπέλα κτλ αρχή της ψηφοφορίας 98. Τέλος. Απορρίπτεται. Πιο γρήγορα σας παρακαλώ να ψηφίζετε. Έχουμε πολλές τροπολογίες. 2. 97. Τροπολογία 97. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 19-22. 99 της κυρίας Χέτ. Ψηφίζουμε 99. Τέλος. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 100 με την προφορική ε, τροπολογία συγγνώμη που βλέπετε. Περ, κατά, εγκρίνεται η προφορική. 100, 101 και τα λοιπά καταπίπτουν. 102 απορρίπτεται. 103 διόν ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 105 αμπάντ. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Καταπιπτήτη 104. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 110. Ψηφίζουμε την 110. Τέλος. Απορρίπτεται. 111. Ψηφίζουμε την 111. Τέλος. Εγκρίθηκε. 22 υπέρ 19 κατά. 112 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 113 ταραμπέλα και τα λοιπά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 116. 116. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 117. Ψηφίζουμε. 117. Τέλος. Εγκρίνεται. 118. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 25 υπέρ 16 κατά. 119. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 120. Ψηφίζουμε την 120. Τέλος. Απορρίπτεται. 14 υπέρ 27 κατά. Συμβιβαστική 18. Ψηφίζουμε. 110. Όχι, συγγνώμη, συμβιβαστική 18 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 24 υπέρ 16 κατά. 124 ντεγιόν ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 3. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 136. Ψηφίζουμε την 136. Τέλος. Απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 140. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 141. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 142. Ψηφίζουμε. Απορρίφθηκε. 143 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 144 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται 145 υπέρ κατά απορρίπτεται 146 υπέρ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 146 τέλος απορρίπτεται επίσης 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Συμβιβαστική 6 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 6 απορρίφθηκε. Έχουμε όλες τις υπόλοιπες λοιπόν που πρέπει να ψηφίσουμε. 116 υπέρ. Α, 160, συγγνώμη. 160 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 159 159 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 161. Τέλος. Απορρίπτεται. 165. Τέλος απορρίφθηκε 162 Α, επιτέλους ψηφίσαμε μία τροπολογία. Την 162. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Συγχαρητήρια. 167. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Η 167 με δύο ψήφους. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Συμβιβαστική 7, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται η συμβιβαστική 7. Θα ψηφίσουμε λοιπόν όλα αυτά και το ΕΛΚ και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι την στήριζαν. Άλλαξαν γνώμη. Η τροπολογία 7 υποστηριζόταν από τέσσερις πολιτικές ομάδες και τελικά μόνο 17 ψήφισαν. Αλλάξατε γνώμη. Ωραία, εντάξει. Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι δεν έγινε λάθος. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Ήθελα απλώς να ξεκαθαρίσω γιατί μόνο 14 υπερψήφισαν αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Αλλάξα τη γνώμη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε την 170. Αρχή της ψηφοφορίας. 170. Τέλος. Απορρίπτεται. 171. Τέλος. Απορρίπτεται. 173. Τέλος. Τέλος. Απορρίπτεται. 177. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 169. Τέλος. Απορρίπτεται. Να δούμε αν θα είστε τυχεροί υπέρ της 168. Κατά. εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε πολύ. Όλες οι υπόλοιπες καταπίπτουν 180. Ψηφίζουμε την 180. Τέλος. Εγκρίθηκε. 181 καταπίπτει. και 182. 183 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 187 του κυρίου Σαμπίνη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά εγκρίνεται. 200 ταραμπέλα και τα λοιπά υπέρ κατά εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Ψηφίζουμε την 10. Τέλος. Εγκρίθηκε. 211 Σαλβίνη υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Δεν ήσταν τόσο κύριε αυτή τη φορά. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 226 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 24 καταπίπτη συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 2.28. Ψηφίζουμε την 228. Τέλος. Απορρίπτεται. 229 ψηφίζουμε. Τέλος, απορρίπτεται. 2.30 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 13, συμβιβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 238 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 2.39 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 246 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 247 ψηφίζουμε την 247. Τέλος απορρίπτεται η 248 καταπίπτει 249 υπέρ κατά υπέρ 249 κατά εγκρίθηκε 250 υπέρ κατά εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά εγκρίθηκε επίσης 251 Αρχή της ψηφοφορίας. 251. Τέλος. Απορρίπτεται. 252. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 261 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 262. Αρχή της ψηφοφορίας. 262. Τέλος. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ παρακαλώ είναι της εισηγήτριας. Κατά. Εγκρίνεται. Τοπολογία 277 ως προστίκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 276 πίπτη. 279. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 279. Πέρασε τη ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 278 υπέρ. Μάλλον ηλεκτρονικά πάλι ψηφίστε. 278. Πέρασε τη ψηφοφορίες. Απορρίπτεται και αυτή. 281. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και 280. Ψηφίστε. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Τροπολογία 282. Σαλντεμόζε υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 284 καταπίπτει. 285 και 286 κρότσμεν συνδυάζονται με την προφορική τοποποίηση. Α, καταπίπτει. Όλες οι άλλες καταπίπτουν. 287 σαλτεμόζα υπέρ, κατά εγκρίνεται, 288 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 289 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 290 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 291 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 293. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 293. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 294. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. 295. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 292 καταπίπτει. 296 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες απορρίπτεται. 297 Ψηφίστε. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες, Απορρίπτεται. 298. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Η ίδια πλειοψηφία. 299. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 301 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 302 υπέρ, ξανά. 302 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 303 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η συμβαστική 19. Θα το λέξουμε όμως ηλεκτρονικά καλύτερα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 33. Υπέρ, παρακαλώ, της 33. Κατά. Απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 35, η γαλλική είναι γλωσσικό, έτσι. Δεν ψηφίζουμε σε αυτό. 36 όμως, 36 τώρα. Υπέρ παρακαλώ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 38, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της ηγήτρες υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 τώρα. Υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Και για τη 44. 42, Απορρίπτεται η 42. 43 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44. Να ελέγξουμε παρακαλώ για τη 44. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ναι, απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 49 υπέρ. Α, εδώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 49. Πέρα στις προφορίες. 20-20 είναι το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται συνεπώς. Τροπολογία 50. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Να ελέγξουμε και εδώ παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. 51. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με διαφορά δύο ψήφους, 18-20. Τροπολογία 52 του κύριου Ντεγιόγκ. Ψηφίστε παρακαλώ για την 52. Απορρίπτεται. 53. Του κυρίου Τεγιόν. Υπέρ παρακαλώ. Για δείξτε με διανατάσεως. Κατά. Απορρίπτεται. 54 του κύριου Τεγιόν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55 Σαλβίνη. Υπέρ. Να ελέγξουμε. 55 Σαλβίνη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 56 του κ. Ντεγιόγκ τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57. Έγκστρομ και άλλων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά εγκρίνεται. 64 64 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 65 υπέρ κατά εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά απορρίπτεται 69 υπέρ κατά απορρίπτεται να ελέγξουμε ωραία 69 ψηφίστε παρακαλώ είναι τροπολογία τύρνα πέρας της ψηφοφορίας είχατε δίκιο εγκρίθηκε με, 60, με 21 ψήφους υπέρ και 19 κατά Τροπολογία 70 Ροσφόρ. Και εδώ ηλεκτρονικά. 70. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71. Δε Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72. Του κύριου Ντεγιόν. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 76 η καταπίπτει. 77 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Ηλεκτρονικά να ελέγξουμε παρακαλώ για την 81. Ψηφίστε. Πέρα στις προφορίες εγκρίνεται. 22-16. Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα 90 καταπίπτει. 92 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Να ελέγξουμε παρακαλώ για την 93. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορία εγκρίνεται με δύο ψήφου διαφορά, λέει ο πρόεδρο. Η επόμενη. κατ 94. 94 τώρα. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροποποιημένη γνωμοδότηση. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 33 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καρχόλα, την απουσία της. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Έχω να κάνω όμως ένα μικρό σχόλιο και μία πρόταση, παρακαλώ. Έχω να κάνω την εξής πρόταση, παρακαλώ, όσον αφορά την ψηφοφορία. Σήμερα θα πρέπει να δούμε την εντολή, την γνωμοδότηση μάλλον μια συναδέλφου για τα οχήματα. Εγώ θα έλεγα να μην ψηφίσουμε σήμερα, γιατί ένα από τα κριτήρια είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και πιστεύω ότι οι θέσεις είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Γι' αυτό προτείνω να μην ψηφίσουμε σήμερα. Μα εδώ πέρα προκαταλαμβάνετε τα πράγματα, λέει ο Πρόεδρο. Ακόμα δεν είχαμε φτάσει εκεί. Δεν ξέρω, οι ο κύριο Παντσέρη δεν είναι εδώ, ε. Ωραία, κάμπ τότε πρώτα. Σίγουρα άκουσα αυτό που είπα ο κύριος Βαντεκάμπ. Θα σας είχα δώσει αλλιώ το λόγο. Κύριε Βαντεκάμπ, Εσεί προτείνετε να σας δώσουμε εντολή με την ομάδα διαπραγμάτευσής σας να πάτε στο Συμβούλιο και να ασχοληθείτε με τον κανονισμό αυτών. Για πείτε μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά την θέση του Κοινοβουλίου που δουλεύει συχνά με δύο αναγνώσεις η πρότασή μου όμως σήμερα είναι να έχουμε μία ανάγνωση. Είναι ένα πολύ τεχνικό ζήτημα αυτό που περιλαμβάνει πάρα πολλές λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα και όλα αυτά τα τεχνικά είναι που έχουμε να εξετάσουμε. Για να επιταχύνουμε λίγο λοιπόν κάπως τη διαδικασία, όπως και ο κύριος Μπαντσέρη, έτσι και εμείς προτείνουμε μία ανάγνωση. Έτσι θα είναι πιο σαφή τα πράγματα για τη βιομηχανία, είναι προτιμότερο για το περιβάλλον και τελικά είναι προτιμότερο και για τη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά, γιατί θα έχει πιο ξεκάθαρες ρυθμίσεις έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πιο ξεκάθαρο κανονισμό. Ο κύριος Κόσνερ είπε ότι δεν έχει οριμάσει ακόμα αρκετά το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Αντιλαμβάνομαι την ε, θέση αυτή, αλλά σύμφωνα με τις δικές μου τις ε, πληροφορίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια αξιολόγηση αντικτύπου. Καλό θα ήταν να έχουμε την αξιολόγηση αυτή αντικτύπου και μετά να πάμε για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θέλει κανείς άλλο το λόγο εδώ, κυρία Κέπαρτ, πριν ψηφίσουμε. Πολύ σύντομα, γιατί θέλουν όλοι να φύγουν. Ενδεχομένω υπάρχει και η ψηφοφορία βεβαίως. Ε. Υπάρχει αν θέλετε, πολύ έντονη κριτική όσον αφορά το κείμενο αυτό και την πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν όμως τεχνικά θέματα, δύσκολα θέματα και εξαιρετικά αν θέλετε θα μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να το ε, πούμε αυτό τώρα. Ο κύριος Βαντεκάπα. Πρόεδρε, μια στιγμή να απαντήσω στον συνάδελφο. Η έκθεση ε, αντικτύπου αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή να μην υπάρχει παρεξήγηση από αυτού. Να μην υπάρχει. Εννοείται ότι πρέπει να την έχουμε. Λέτε λοιπόν ότι θα ληφθεί υπόψη αυτή η έκθεση αντικτύπου, έτσι κι αλλιώς. Ωραία η κυρία Και εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ. Μπορούμε να πείσουμε, πιστεύουμε, το Συμβούλιο. Το θέμα είναι βεβαίως ότι δεν μπορούμε βάσει των ε, ισχύουσων ε, διατάξεων σήμερα να συμφωνήσουμε πριν από την πρώτη ανάωση με το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να βρεθεί συμβιβασμός. Εάν όχι, θα πάμε όπως προβλέπει η διαδικασία στην Ολομέλεια. Μια και δεν είναι εδώ ο θα μιλήσετε εκ μέρους του. Κύριε Γκέπχαρτ για τους ελκυστήρες. Μα εγώ μίλησα για τον εκ μέρους του κύριου Παντσέρη. Το έκανα ήδη. Εντάξει, τότε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τις δύο προτάσεις. 21 ψήφους υπέρ χρειαζόμαστε. Ας ψηφίσουμε ξεχωριστά. Πρώτη ψηφοφορία. Ναι ή όχι, ξεκινάμε τώρα διαπραγματεύσεις για τα οχήματα. The vote's closed. Τέλος. 19 υπέρ 3 κατά. Άρα δεν είναι εντολή σήμερα. Δεν υπάρχει εντολή, δεν είναι αρκετή. Θα ψηφίσουμε για τα... Για τους ελκυστήρες τώρα. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για τους ελκυστήρες. 23 υπέρ. Ωραία. Έχετε την εντολή, ο κύριος Παντζέρη μάλλον έχει την εντολή για τους ελκυστήρες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα. Κύριε Μπίλαν, ε, κύριε Ροσφόρα, η έκθεση κυρίας Κόρολα πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Έχουμε την Επιτροπή όσον αφορά βεβαίως τη μελέτη αντικτύπου για τις προτάσεις σας. Θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο. Κύριε Μπίλαν, καταρχήν, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη συζήτηση βεβαίως. Και δεδομένου ότι έχουμε την Επιτροπή για τη μελέτη αντικτύπου, θέλετε να ξεκινήσει η συζήτηση για την έκθεσή σας και κατόπιν θα βρούμε χρόνο αργότερα μεταξύ ημών και των σκιωδών εισηγητών σε μια άλλη συνεδρίαση. Έχουμε μισή ώρα και μπορούμε να την αφιερώσουμε κατόπιν στην έκθεση του κυρίου Ροσφόρ, πρόγραμμα καταναλωτές. Ξέρω ότι δεν είναι ικανοποιητική αυτή η λύση που σας προτείνω, αλλά δεν βλέπω άλλη. Αυτό σημαίνει ότι θα αναβάλουμε βεβαίως και την ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών που αρχικά έχει προβλεφθεί για τις 28 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Έτσι και δεν βλέπω πολλούς από τους σκιώδεις παρόντες. Κυρία Σαμπρίζ δεν είναι εδώ, Σάλτερ Μόζερ δεν είναι. Λόκεγκαρντ επίσης, λείπει. Α, όχι είναι. Η κυρία Ρουλέ είναι εδώ. Σαλβίνη λείπει. Άρα, αφού λείπουν οι σκιώδεις, οι περισσότεροι, μου φαίνεται ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια στιγμή με τους σκιώδες να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να συζητηθούν και οι τροπολογίες και κατόπιν να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Ε, σε αυτή την περίπτωση να αναβληθεί όλη η συζήτηση. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, αλλά θα πρέπει, και το ζητώ από τους ε, συντονιστές, να είναι παρόντες την επόμενη φορά όλοι οι σκιώδεις. Γιατί να μην ξεκινήσουμε. Κάντε μας την παρουσίασή σας. Κάντε μας την παρουσίαση της πρότασής σας, κύριε Μπίδε. E, e, το σύστημα IMI που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών επί τη βάση της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών ιδιωτήτων λειτουργεί μετά από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς δεν έχουμε κάποιο νομικό μέσο σαν βάση για αυτό και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για τη διεύρυνση της χρήσης του συστήματος. Είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την ε, καθημερινή συνεργασία ανάμεσα στις διοικήσεις των κρατών μελών, τις δημόσιες διοικήσεις και ε, βοηθά γενικά να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται πολλές φορές. Ε, πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια τακτική θα έλεγα νομική διαδικασία και η πρόταση ενοποιεί όλα τα στοιχεία του συστήματος σε ένα μεμονωμένο νομοθετικό μέσο. Αν πρέπει να διευρυνθεί όμως το μέσο αυτό και σε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αυτό θα πρέπει να γίνει επί τη βάση νέων κανονισμών. Δεν συμπεριλαμβάνω εδώ τις κατεξουσιοδότηση ε, πράξης. Η διεύρυνση λοιπόν του συστήματος IMI θα απαιτήσει στο μέλλον να υπάρξουν κάποιες αλλαγές του συστήματος ενημέρωσης ε, για την εσωτερική αγορά που είχε αποφασιστεί στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα της αποθήκευσης δεδομένων, άρθρο 13. Εκεί εισάγεται η ανάγκη για τη διατήρηση και αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Έξι μήνες ε, είναι τώρα. Δεν έχουμε μελέτες επιπτώσεων για τη συγκεκριμένη αυτή πρόβλεψη και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω να εμείνουμε στις υπάρχουσες λύσεις σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων. Και το τρίτο θέμα είναι η προσβασιμότητα προς τρίτους, εξωτερικούς και μη. Η σωστή λειτουργία του MIMI, IMI ε, μάλλον είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Αλλά από την άλλη θα πρέπει το σύστημα αυτό να μην ανοίγει προς τρίτους αν δεν έχει υπάρξει μια μελέτη των επιπτώσεων μιας τέτοιας μορφής συνεργασίας λεπτομερείς συζητήσεις δεν έχουν γίνει ακόμα, θα πρέπει να ξεκινήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μια συνάντηση, είχαμε μια συνάντηση με την Προεδρία, με τους δύο σκιώδεις συζητητές και θα οργανωθούν περαιτέρω συναντήσεις στο μέλλον. Να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους. Είμαι δεκτικό σε κάθε τροπολογία μέσω της οποίας μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική και κοινά αποδεκτή λύση, γιατί η σωστή λειτουργία του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά είναι κάτι το πολύ θετικό για την ίδια την αγορά και διευκολύνει τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Παρβάνοβα, Ρούλε και Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπίλαν. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα η συγγήτρια και γι' αυτό μου ζήτησε να μεταφέρω τις ιδέες της γύρω από την έκθεση Μπέλαν. Η έκθεση Μπέλαν είναι μια πρόταση η οποία νομίζω δεν θα ενισχύσει τελικά, δεν θα καταστήσει πιο ισχυρή την Νομίζω ότι η συνεργασία στον τομέα της μετακίνησης και της κινητικότητας καλύτερα των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων κτλ. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ και απαιτείται διοικητική θα έλεγα ευκρίνεια έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς χρειάζεται για να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον. Συνεπώς δεν θα υποστηρίξω την πρόταση του κυρίου Μπέλαν. Ε, θα θέλαμε εμείς να επιστρέψουμε στην αρχική ιδέα που ήταν η ιδέα της διοικητικής συνεργασίας. Δεύτερον, και εμείς κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο ο κύριος Μπίλαν θέλησε να μην υπάρχει συνεργασία με τρίτους γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα ως εκ τούτου είναι κατανοητό να μην υπάρχει άμεση κυκλοφορία τους. Από την άλλη όμως το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι εθνικές αρχές να μπορούν να παρεμβαίνουν και θα πρέπει οι εθνικές αρχές να είναι σε θέση να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις επιθυμίες τους σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια συνένεση, ότι δεν θέλουμε δηλαδή να συμπεριληφθούν. Μπορούμε εδώ να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το θέμα είναι πότε τα δεδομένα αυτά θα σβήνονται σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρατείνει την προθεσμία διατήρησης. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στη σωστή λύση όμως και πώς η προστασία των δεδομένων θα παίξει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Τα θέματα του απορρίτου ή τα θέματα καλύτερα της εμπιστευτικότητας, αυτά είναι βασικά θέματα και κάποια από τα δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται μερικές φορές θα εξάγονται σε εισαγωγικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην απασχολήσει. Το σύστημα πρέπει να είναι λειτουργικό, πρέπει να είναι ασφαλές, πρέπει να είναι τυχή, ταχύ εφόσον θέλουμε η οδηγία αμοιβαία αναγνώρισης πτυχίων κτλ να είναι αποτελεσματική έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ για την καταγραφή αυτών των δεδομένων, να εντοπίσει σωστά τα προβλήματα και έτσι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία να έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με τον σωστό τρόπο. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ πρότεινε να γίνει μια δοκιμή όσον αφορά την αντοχή αυτού του όλου συστήματος. Και πιστεύω ότι αυτή η αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να προχωρήσει με τις απαραίτητες εγγύησεις και δικλείδες ασφαλείας. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρντ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος ε, της ε, σκιώδους εισηγήτριάς μας, δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα, και εξ ονόματός της θα ήθελα να πω ότι και εμείς υποστηρίζουμε αυτήν την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής θεωρούμε ότι σαφώς ε, θα μπορέσει να αποτελέσει μια σωστή νομική βάση ε, αυξάνοντας τη νομική ασφάλεια, κάτι το οποίο σαφώς χαιρετίζουμε ή θα μπορούμε να εργαστούμε πολύ καλύτερα. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο προϋποθέτει ότι πολλοί τομείς θα παραμείνουν ακόμα ανοιχτοί. Είδα τις τροπολογίες του κυρίου Βίλαντ δεν θεωρώ ότι όλες οι προτάσεις αυτές είναι καλές. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε όλες τις δυνατότητες ε, ελιγμού. Επαναλαμβάνω, κάποιοι τομείς θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Η προστασία των δεδομένων είναι παραδείγματος χάρη ένας πολύ σημαντικός ε, τομέας. Η εξωτερική πρόσβαση, μάλλον η πρόσβαση τρίτων σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να ε, εξεταστεί πολύ προσεκτικά ποιος έχει πρόσβαση. Εδώ υπάρχει και άλλη μια τροπολογία του κυρίου Βίλαν. Δεν πρέπει να περιορίσουμε υπερβολικά την πρόσβαση, αλλά βεβαίως η προστασία των δεδομένων είναι εδώ καθοριστική. Όχι μόνο όσον αφορά την αποθήκευση των δεδομένων, αλλά και του χρόνου, της διάρκειας ε, αποθήκευσης τους. Πόσο καιρό μπορεί κανείς δηλαδή να διατηρήσει κάποια δεδομένα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Θεωρώ όμως ότι πραγματικά η υποβολή αυτών των προτάσεων είναι κάτι που το περιμέναμε εδώ και χρόνια και επιτέλους θα τεθεί μια νομική βάση και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παντάνοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του σκιώδους του κυρίου Λόκιγκαρτ και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω την γνωμοδότησή του. Καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Μπίλαν για την εργασία που έχει κάνει για το θέμα αυτό. Είναι δύσκολο το θέμα και ο κύριος Λόκιγκαρτ θεωρεί ότι είναι πολύ καλή η προσπάθεια, έχει παρόλα αυτά κάποια σχόδια. Όσον αφορά την διοικητική συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό είναι κάτι που όπως προτείνει ο κύριος Μπίλαν πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεργασία βάση του συστήματος ε, του Ευρωπαϊκού IMI, περισσότερη λοιπόν ε, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία και βεβαίως αυτό επεκτείνεται και σε άλλα δεδομένα αλλά και στην ε, αμοιβαία αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων και των διπλωμάτων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στα παραρτήματα 1 και 2 που ιδιαίτερα στο παράρτημα 1 αναφέρεται η πιθανή εφαρμογή του IMI και σε άλλους τομείς. Όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, ο κύριος Λόκεγκερ θα ήθελε αυτή η πρόταση να εξεταστεί περισσότερο ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις. Επίσης, όσον αφορά την αποθήκευση των δεδομένων. Έξι μήνες είναι η διάρκεια αποθήκευσης. Η πρώτη σου εισηγητή είναι να πάμε στους 13 μήνες. Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία, θεωρεί ο κύριος Λίκεγκαρτ. Αλλά όσον αφορά την μεγαλύτερη διάρκεια για την φύλαξη των δεδομένων θα πρέπει να κοιτάξουμε και σε άλλες οδηγίες τι προτείνεται, τι διάρκεια υπάρχει την ίδια ώρα. Εδώ δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Υπάρχει ε, σαφώς και η περίπτωση εξέτασης εσφαλμένων δεδομένων και διόρθωσή τους. Επίσης, η πρόσβαση σε εξωτερικούς ε, φορείς. Ναι, βεβαίως περισσότερη ευελιξία για την εσωτερική χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος και σε άλλους τομείς του συστήματος IMI. Παρ' όλα αυτά, ο κ. θεωρεί ότι η εξωτερική φορείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ατόμων ή εμπιστευτικά ή απόρριτα δεδομένα επιχειρήσεων. Η ε, κυρία Ρίλε. Χαίρομαι γιατί εγώ δεν χρειάζεται να διαβάσω το χαρτί κάποιου άλλου. Είμαι προσωπικά εδώ και μπορώ να μιλήσω για ε, τον εαυτό μου. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτάσεις που κάνει. Υπάρχουν σημεία με τα οποία διαφωνούμε όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, ιδιαίτερα πρόσβαση εξωτερικών φορέων ή τρίτων. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ανοίξει αυτό το σύστημα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγγύσεις και γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Μπίλαν θέτει το θέμα αυτό Αυτά βέβαια που προτείνει ουσιαστικά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να βρούμε διαφορετικές λύσεις για την κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φύλαξη των δεδομένων, την αποθήκευση και την καταστροφή τους. Ευχαριστώ πολύ. Good. Well, thank you all very much, um, acting Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον εισηγητή από την Επιτροπή. Θέλετε να μας ε, κάνετε κάποια σχόλια, μας πείτε ποιος είσαστε και πολύ σύντομα να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Από αυτή την πλευρά χαιρόμαστε που βλέπουμε γενική στήριξη και από τον κύριο Μπίλεν αλλά και από τους σκιώδεις εισηγητές. Οι δικές μας ανησυχίε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναφέρθηκαν και από τους ομιλητές εδώ. Θέλουμε να διατηρήσουμε το πεδίο εφαρμογή στην διοικητική συνεργασία και όχι μόνο στην ανταλλαγή πληροφοριών. Όσον αφορά τώρα τους εξωτερικούς ε, φορείς, όπως υπόθηκε η και είναι ζωτικής σημασίας για το Solvit, όταν υπάρχουν ε, ε, προσφυγές από τους πολίτες. Θέλουμε λοιπόν να, διατηρηθούμε, να διατηρήσουμε μάλλον τους εξωτερικούς φορείς εντελώς χωριστά από το IMI. Όσον αφορά τώρα το μηχανισμό επέκτασης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις κατεξιζότητες πράξεις, την πρόταση δηλαδή για αυτές, αλλά αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ είναι η εξαφάνιση πειραματικών ε, σχεδίων. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε δοκιμές, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό θέλουμε να διατηρηθούν. Για τον χρόνο πριν την ε, διαγραφή των στοιχείων, η πρώτη επιτροπή στη ότι τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται το πολύ για 18 μήνες. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις θα έχουν διαγραφεί πολύ νωρίτερα. Και ακόμα και σήμερα έχουμε για τις υπηρεσίες προσωπικά δεδομένα ε, το οποία δεν κρατάμε καθόλου. Δηλαδή τα κλείνουμε αμέσω, σε μηδέν χρόνο τα κρατάμε. Αυτό που θέλουμε εδώ να πούμε είναι ότι μένουμε στις περιόδους εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα ε, για την δουλειά που κάνουμε, για το Solvit. Είναι τρία χρόνια η περίοδος αυτή. Οπότε ήδη οι 18 μήνες είναι μείωση. Τους χρειαζόμαστε τους 18 μήνες. Γιατί συχνά άνθρωποι των οποίων το πρόβλημα έχει λυθεί μέσω του Solvit μετέρχονται σε εμά γιατί διαπιστώνουν ότι δεν ε, τίθεται σε εφαρμογή η λύση. Γι' αυτό καλό είναι να μπορούμε στην βάση δεδομένων να τα ξαναβρούμε τα στοιχεία τους και αντί να τους λέμε ότι α, διαγραφήκανε τα δεδομένα αυτά οπότε αυτού και από την αρχή. Συνεπώς αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που είχα και φυσικά και ευχαρίστω θα συνεργαστούμε και με τον εισηγητή και με τους σκιώδες. Και ελπίζω να υπάρξει περαιτέρω πρόεδρο στο θέμα αυτό. Κύριε Μπίλαν, θέλετε να συνοψίσετε. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως θα προσπαθήσω να κάνω την σύνοψη των όσων άκουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν σύντομη η συζήτηση σήμερα. Δεν είχαμε χρόνο για περισσότερη επεξεργασία του θέματος. Βεβαίως από εδώ και πέρα χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρινήσεις που περιμένουμε να μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φάνηκαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αυτό ίσως δεν θα ήταν τόσο εμφανές αν από την αρχή είχαμε τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου από μέρους της Επιτροπής. Η πρόταση της Επιτροπής είναι ουσιαστικά μία κωδικοποίηση του status quo. Δεν αλλάζει τίποτα. Αν κοιτάξουμε λοιπόν το πώς προστατεύονται σήμερα τα προσωπικά δεδομένα, εγώ θα πρότεινα να παραμείνουμε στην ε, υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την διάρκεια φύλαξης. Λαμβάνω υπόψη μου τον επιθεωρητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τις ανησυχίες που έχει εκφράσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ωραία, θα δούμε τι θα οργανώσουμε για την συνάντηση που πρέπει να λάβει χώρα με τους σκιώδεις Αν χρειάζεστε και άλλη δημόσια συζήτηση, φυσικά και θα την οργανώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και την Επιτροπή και θα προχωρήσουμε στο τελευταίο μας σημείο που είναι το πρόγραμμα καταναλωτές για την περίοδο 2014-2020. Η κυρία Μάια θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Βεβαίως ε, θα ακούσουμε και σχόλια και ενδεχομένως ε, ερωτήσεις αν υπάρχουν θέλετε να παρουσιάσετε εσείς ή να δώσετε το λόγο στην κυρία Μάινχαρτ. Euh, Πρόεδρε, ευχαρίστω. Αν έχουμε μισή ώρα για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα, ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια θα πρέπει να είναι σύντομη, γιατί αλλιώς θα αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει και μετά να ανταλλάξουμε απόψεις στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Δεν θέλω όμως να το σφάξουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το θέμα. Έτσι στα γρήγορα. Έχουμε μιλήσει με τους διερμηνείς και θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο παραπάνω. Ας πούμε ότι έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας. Το κεντρικό θέμα πάντως θα είναι η παρουσίαση της κυρίας Μάινερς. Αυτό θα είναι το βασικό. Οπότε Σάκη Μάινεν, που είναι γενική διευθύντρια για τι ε, του καταναλωτή. Κύριε Ταραμπέλα, α, μετά έχετε θέλετε το λόγο. Εντάξει, παρακαλώ κύριε Μάινερ. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δύο εισαγωγικέ παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα Σήμερα σας παρουσιάζω το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020. Μετά το τρέχον πρόγραμμα, το οποίο λύγει το 2013 και συνοδεύει βέβαια και την ατζέντα για τους καταναλωτές που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ο, και σχετικά με την οποία την Πέμπτη θα έχουμε ακρόση. Δεν λέω ότι το ένα συνδυάζεται απόλυτα με το άλλο, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι ανταλαμβανόμαστε ότι το πρόγραμμα στηρίζει την ατζέντα και ότι η ατζέντα αναφέρεται στο πρόγραμμα. Το πρώτο που θα σας πω είναι τεχνικό αλλά πολύ σύντομα είναι με τη μορφή κανονισμού η πρόταση. Το τρέχον πρόγραμμα είναι απόφαση. Αυτό όμω δεν είναι καμιά ιδιαίτερη διαφορά και γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση, εάν υπάρχουν ε, άμεσα ωφέλη σε διάφορες οργανώσεις, τότε θα πρέπει να μιλάμε για κανονισμό και επειδή έχουμε και άλλα προγράμματα ε, βάση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, όλα αυτά είναι κανονισμός και για να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει συνοχή. Τώρα όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών. Ποιοι είναι οι στόχοι, αναφέρονται εδώ πέρα, τους βλέπετε. Το πρόγραμμα βασίζεται σε πολλές πηγές. Βασίζεται στην μεσοπρόθεσμη εξολόγηση του τρέχοντος προγράμματος και σε μια έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου που έχετε στη διάθεσή σας. Είναι κάτι που συζητήσαμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και με τα μέλη του δικτύου για την πολιτική για τους καταναλωτές, με υπουργεία, με οργανώσεις καταναλωτών και λάβαμε επίσης υπόψη μας και διάφορες εκθέσεις που έχετε εσείς ετοιμάσει η Επιτροπή σας, Σάλτε Μόζα, και άλλες. Η πολιτική για τους καταναλωτές είναι σχετικά νέα σε ηλικία. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε νέες προκλήσεις. Θα διαπιστώσετε όμως παρόλα αυτό ότι υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στο τρέχον πρόγραμμα και το προτινόμενο μελλοντικό πρόγραμμα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε υπό το φως της αξιολόγησής μας είναι να λάβουμε υπόψη μας τις δαπάνες και να τις ξαναδούμε ανάλογα με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά λοιπόν το συνολικό προπολογισμό, είναι ένα συνολικό προπολογισμό 197 εκατομμυρίων ευρώ για 7 χρόνια, 2014 με 2020, που σημαίνει 175 σε τιμές του 2011. Πρόκειται για μια πολύ μικρή αύξηση σε σχέση, σε σχέση με τις τρέχουσες δαπάνες το τρέχον πρόγραμμα και περιλαμβάνει και τις διοικητικές δαπάνες. Για παράδειγμα, οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τους εκτελεστικούς οργανισμούς που χειρίζονται τον προπολογισμό. Συνεπώς, δημοσιονομικά είναι ένα μικρό πρόγραμμα. Αξίζει όμω τον κόπο να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποφάσισε να διατηρήσει το τρέχον επίπεδο δαπανών παρά ε, τη, τους περιορισμούς που υποβάλλονται γενικότερα στα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα. Έτσι καλώς είναι σταγόνων το κενό. Προσπαθούμε να βάλουμε χρήματα εκεί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια διαφορά. Βιάστηκα, πήγαινε πίσω παρακαλώ στην προηγούμενη. Λοιπόν, κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε στην υπάρχουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα δηλαδή για τους καταναλωτές φροντίζει για δαπάνες στο RAPEX που είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για προϊόντα επικίνδυνα για τον καταναλωτή. Έπειτα θέλουμε ε, να δώσουμε χρήματα για δράσεις οι οποίες έχουν νόημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πράξεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Στηρίζουμε για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών που στηρίζει τους καταναλωτές που έχουν προβλήματα με αγορές που έχουν κάνει διασυνοριακά. Επίσης βάζουμε χρήματα για να συλλέξουμε στοιχεία, για να έχουμε δηλαδή μια βάση δεδομένων όσον αφορά ε, τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στηρίζουμε και σε ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών. Τρίτον, στηρίζουμε και εθνικές δράσεις, εθνικές πρωτοβουλίες, προκειμένου αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ή ακόμα και διοικητική ενίσχυση. Τώρα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν τέσσερις ειδικοί στόχοι με ανάλυση προσωρινή καταρχήν των δαπανών. Έχουμε ασφάλεια, κάπου 22% του προπολογισμού, ενημέρωση και κατάρτιση, που είναι στήριξη οργανώσεων καταναλωτών είναι ε, δικαιώματα και διόρθωση, επανόρθωση και είναι και η ε, τήρηση και η εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Εποφελούνται διάφορες ε, αρχές, Ευρω... τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, πλατφόρμες σε ευρωπαϊκά επίπεδα κλπ. Τώρα τι αλλαγές έχουμε σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα. Το επόμενο πρόγραμμα επικεντρώνεται περισσότερο στην, ε, στις δαπάνες για την εφαρμογή των κανόνων για την τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και όλων των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα τίθεται σε εφαρμογή στην πράξη. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε πρόκειται για τα δικαιώματα των καταναλωτών κάτι το οποίο ενισχύεται και μέσα από το δίκτυο των Εθνικών Αρχών Επιβολής. Μιλάμε ε, για μια αύξηση δόση χρηματοδότησης σε 70% και 50% που ήταν. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, πιστεύουμε για την επανόρθωση. Εδώ φτιάχνουμε την πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών online. Υπάρχει μια πρόταση επιτροπής που βρίσκεται προς εξέταση στην επιτροπή σας. Και τέλος, ξανα... Μάλλον εξυγχρονίζουμε κατά κάποιο τρόπο και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την διαπαιδαγώγηση. Ε, για να ανταποκρινόμαστε περισσότερο στις ανάγκες του 21ου αιώνα και όχι του 20ου. Έχουμε δηλαδή μια πιο διαδραστική φόρμουλα. Δουλεύουμε με δασκάλους και άλλους παιδαγωγούς. Προσπαθώ να πάω γρήγορα και ελπίζω να σας έδωσα κάποια στοιχεία για να σχολιάσετε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσει η συζήτηση από πλευράς μας, έχουμε λίγο χρόνο. Ο εισηγητής. Δεν ξέρω αν ο κύριος Φαμπ θα θέλει το λόγο, ο κύριος Μπούσετλ δεν είναι εδώ. κυρία Ρούλε θα θέλει το λόγο, θα δούμε. Και ο κύριος Ταραμπέλα επίσης έχει ήδη πει. κύριος έχει το λόγο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα τα πω λίγο βιαστικά. Δύο πράγματα πρέπει να μας ικανοποιήσουν. Πρώτον, ότι η έκθεση ανταποκρίνεται σε αυτό που είχαμε ζητήσει πριν λίγα χρόνια. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα καταναλωτές που ε, είναι αποδεσμευμένο από το πρόγραμμα για την υγεία. Δεύτερον, υπάρχει ένας προϋπολογισμός, όχι ιδιαίτερα ισχυρός, αλλά στέκει εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και δεν θα διαμαρτυρηθώ γιατί μειώθηκε ακόμα περισσότερο η εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, εξέφασε το παράδοξο ότι δηλαδή το Consumer Agenda θα έρθει σε συζήτηση μετά από το Consumer Program. Η ατζέντα του καταναλωτή θα έχει μεγαλύτερο εύρος και θα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες θα είναι πιο δεσμευτικές και για άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής. Από την άλλη βέβαια έχουμε να κάνουμε με κάτι ανάποδο από αυτό το οποίο κάνουμε συνήθως. Ελπίζω αυτό να μην έχει αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Μια γενική παρατήρηση παρόλα αυτά. Ο προϋπολογισμός όπως είπα διατηρείται. Παρόλα αυτά έχουμε να κάνουμε ε, με κάτι το οποίο βάζει την κατανάλωση στο κέντρο της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής και τον καταναλωτή στο κέντρο της πολιτικής. και ίσως σε ένα από τα κάνω ένα υπολογισμό και βλέπω ότι με 5 εκατομμύρια κατέτος σε σταθερές τιμές σημαίνει ότι δίδουμε 5 σαντίμ, 5 ε, ε, λεπτά ε, ε, ανακαταναλωτή. Αυτό δείχνει ότι τα χρήματα είναι λίγα και δεν πρέπει να τα χάσουμε γιατί κινδυνεύουν αυτά τα λίγα να μην είναι και αποτελεσματικά. Πρέπει να το σημειώσουμε. Αυτό που με στεναχωρεί σε επίπεδο γενικών παρατηρήσεων είναι ότι καλό είναι που διατηρεί κανείς αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη με ένα τόσο μικρό ποσό. Από την άλλη όμως διερωτώμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά ανοιχτή στις νέες προκλήσεις. Η παράταση των ισιών των προγραμμάτων δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά υπάρχει η κρίση, ο καταναλωτής ε, είναι εύθραυστος, η ενιαία ψηφιακή αγορά δημιουργείται σιγά σιγά, γυράσκει ο πληθυσμός η παγκοσμιοποίηση της κατανάλωσης, όλα αυτά θα έλεγα δεν έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τους στόχους. Sur 1, alors là, euh, moi comme Madame Minor, je Όπως και η κυρία Μάινο χαίρομαι, χαίρομαι διότι πράγματι ειδικά για το ΡΑΠΕΞ υπάρχει μια σαφής βελτίωση υπάρχει ένας προϋπολογισμός που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό του ΡΑΠΕΞ. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης το άνοιγμα του ΡΑΠΕΞ σε όλες τις χώρες είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και να μην ξεχνάμε ιδιαίτερα με την Κίνα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, θα έλεγα σημειώσεις ε, σχετικά με προϊόντα από την Κίνα που παρουσιάζουν κινδύνους στην κατανάλωση για τον δεύτερο στόχο, δηλαδή ενημέρωση και εκπαίδευση του καναλωτή. Εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πριν είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις των καταναλωτών και των ευρωπαϊκών ονόσεων καταναλωτών. Ε, διευκρινίζω ότι ε, όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή για το συνολικό πακέτο ε, αναφέρονται στη συγκεκριμένη διατύπωση. Δίνεται η δυνατότητα μέσω του προγράμματος ΤΡΑΣ στις εθνικές οργανώσεις των καταναλωτών να εκφράζονται. Βέβαια τα χρήματα τα οποία τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών ποικίλουν ανάλογα με το κράτος μέλος. Λυπάμαι γιατί μιλάμε πάρα πολύ για νέους και ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται διαβίου κατάρτιση. Την ξεχνάμε αυτή. Με ενδιαφέρει όμως το ότι προχωράμε στα πλαίσια της διαφάνειας των αγορών ενώ θα ήθελα να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτά που ονομάζω το πιστότοπι σύγκρισης. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές. Να πω επίσης ότι οι επιχειρήσεις ε, θα έχουν να κερδίσουν πολλά από το πρόγραμμα των καταναλωτών. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν ε, θα έλεγα είναι ιδιαίτερα φιλικές προς τον καταναλωτή, δεν ενημερώνουν σωστά τον καταναλωτή γιατί το δίκαιο του καταναλωτή είναι πάρα πολύ περίπλοκο αλλά και για τις επιχειρήσεις είναι περίπλοκο. Ο τρίτος ε, στόχος αφορά τις δυνατότητες ε, προσφυγής, αμφισβήτησης, αποζημίωσης κτλ. Τα συστήματα τα οποία προβλέπονται είναι ικανοποιητικά. Σε σχέση με τις εναλλακτικές διευθετήσεις υπάρχουν σε άλλες τομές, σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς μάλλον, αλλά δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκούν. Ε, για το τέταρτο τώρα, για το σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι πάρα πολύ θετικό να υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης να περάσει από το 50% σε 70%. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε χώρες όπου δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα να προχωρήσουν. Θα ήθελα και το ξέρει αυτό η Επιτροπή να, μου, να πει ότι όταν αυξάνεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγα, διαφάνεια σε αυτά τα κέντρα του καταναλωτή. Γιατί μόνο 15% των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν τη λειτουργία των κέντρων αυτών και πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Λοιπόν, αυτά ήθελα από σαν εισηγητής. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα εμπλουτίσουν την συζήτηση αυτή ε, με μεγάλη ταχύτητα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν αφήσατε και πάρα πολύ χρόνο για τους συναδέλφους σας, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να δώσουμε και το χρόνο στην κυρία Μάνα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για την αρχή της διαδικασίας. Η κυρία Περές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πράγματι σύντομη. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσίασή της για το νέο αυτό πρόγραμμα που είναι ζωτική σημασία για να διασφαλίσει μια εσωτερική αγορά πιο δυναμική και πιο ανταγωνιστική. Πράγματι, αν θέλουμε ο καταναλωτής να αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης, τότε πρέπει οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά, να είναι πρωταγωνιστές μέσα σε αυτή την αγορά και άρα να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και να είναι καλά προστατευμένοι. Στην περίπτωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών διασυνοριακά πρέπει να είναι πολύ προστατευμένη. Δεύτερον, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών από τη μία και από την άλλη μεριά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Προς το παρόν φαίνεται ότι η εσωτερική αγορά προχωράει πιο γρήγορα από την προστασία των καταναλωτών. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη φορά θέλει να ενισχύσει τον ρόλο των οργανώσεων των καταναλωτών για να μπορούν πράγματι να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και στην ενημέρωση αλλά και στη στήριξη των καταναλωτών και για να ε, υπάρχει μια πλατφόρμα ε, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από όπου να μπορεί να αποφεληθεί ο καταναλωτής. Θέλω επίση να υπογραμμίσω και ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι δεν υπάρχει αρκετά στο νέο αυτό πρόγραμμα. Πρόκειται για την προστασία μιας ειδική καταγορία ευάλωτων καταναλωτών. Βέβαια, είναι φιλόδοξη η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλα αυτά, ο κανονισμός δεν λέει ότι το πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αύξηση των ευάλωτων καταναλωτών και την ε, ειδική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και που κινδυνεύουν μερικές φορές να βρεθούν στο περιθώριο. Εγώ θα ήθελα να δω ειδικέ δράσεις υπέρ αυτών των ευάλωτων καταναλωτών γιατί έτσι θα μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική προστασία όλων των καταναλωτών. Όταν κάποιος είναι ευάλωτος ως καταναλωτής, δεν τολμάει καν να αγοράσει, δεν καταλαβαίνει την ενημέρωση έτσι όπως του φτάνει και δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του, πώς θα αποζημιωθεί, πώς θα ζητήσει επανόρθωση. Γι' αυτό λέω ότι θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί και στα ηλικιωμένα άτομα και στους ευάλωτες καταναλωτές. Σίγουρα δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι είναι και πολλοί άλλοι ευάλωτοι καταναλωτές. Ευχαριστώ. Κύριε Ταραβέλα, είχατε πει ότι θέλατε και εσείς το λόγο. Ε? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω πραγματικά ότι λείπει ενθουσιασμός, λείπει πάθος, λείπει φιλοδοξία από τις προτάσεις αυτές. Ουσιαστικά γίνεται αναφορά στο RAPEX. Βεβαίως και χρειάζεται βελτίωση των δυνατοτήτων του συστήματος αυτού. Θα ήθελα να αναφέρω πέντε σημεία. Πρώτον, στο κέντρο θέλουμε να βάλουμε τον καταναλωτή. Ουσιαστικά όμως δεν κάνουμε απολύτω καμία πρωτοβουλία έτσι ώστε αυτή η ιδέα να ενσωματωθεί ε, εκεί που είχε ενσωματωθεί και σε δύο άλλες οδηγίες όσον αφορά την ε, πίστη, την τελειωτική δυνατότητα και τη δυνατότητα να γίνουν μελέτες για να δούμε τις επιπτώσεις. Δεύτερο σημείο, ενημέρωση του καταναλωτή. Μια σημαντική προτεραιότητα, χωρίς όμως να έχουμε μέσα ο προϋπολογισμός. Μας επιτρέπει να κάνουμε μία έρευνα πολυσέλιδη, 376 σελίδες, που μας δίνει στοιχεία για το 2011-2012. Είναι, κατά την άποψή μου, άχρηστες αυτές οι μελέτες και θα πρέπει να μην επαναλαμβάνονται στο μέλλον. Όσον αφορά το scoreboard, αυτό το βαθμολόγιο, συμφωνώ με τον Ρομπέρο Σφόρτ. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά πλήττουν τους πιο ευάλωτους. Και το Συμβούλιο Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών δείχνει σήμερα ότι θα πρέπει να επεκταθούν αυτές οι πρωτοβουλίες και σε άλλες ε, περιοχές και σε άλλα κέντρα, τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε και να προβάλλουμε. Τέταρτο σημείο ενημέρωση των καταναλωτών. Έχουμε καταναλώσει 9 εκατομμύρια ευρώ. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. 9 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση των καταναλωτών, πρόγραμμα Ντολτσέτα. Μεγάλη αποτυχία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα σε κάποιες χώρες σχολές για την κατανάλωση, για τους καταναλωτές και θα πρέπει ίσως να διδαχθούμε από τα αποτελέσματα αυτών των σχολών. Πέμπτο σημείο, η Επιτροπή λέει ότι θα συνεισφέρει στην στρατηγική 2014-2020. Δεν βλέπω όμως καμία απολύτως πρωτοβουλία η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, του ηλικιωμένου και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για μια πιο ορθολογική κατανάλωση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στους στόχους μας. Θα πρέπει να σταματήσουμε τις σπατάλες και να γίνει καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων. Για το 2014-2020 κάποιες επενδύσεις, κάποιες δαπάνες θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση. 25 εκατομμύρια έλεγε ο Ρομπέρο Σουό, δηλαδή 5 cents ανά κάτοικο. 0,0002% ουσιαστικά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Περί αυτού πρόκειται. Έχουμε δύο λεπτά για τους εισηγητές και θα δούμε πότε θα μπορέσουμε να πάρουμε τις απαντήσεις από μέρους Επιτροπής αργότερα. Α, κύριο Σφάπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, για τα προγράμματα αυτά, μπορούμε σαφώς και να συζητήσουμε την ατζέντα και να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας καλύτερα αυτούς τους πόρους. Περισσότερα βεβαίως θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να κάνουμε. Βλέπουμε όμω ότι τα μέσα που μας δίνει αυτός ο προεμβολιό μου είναι πολύ περιορισμένα και ελπίζω η Επιτροπή στην επόμενη πρότασή τη να μας προτείνει κάτι περισσότερο. Δεύτερον, ο ρόλος των κέντρων προστασίας του καταναλωτή, ο οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί. Η συγχρηματοδότηση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα μόνο για τα νέα κράτη-μέλη. Για τα παλιά κρατημέλη δεν είναι πρόβλημα. Τα νέα κρατημέλη μας λένε γιατί θα πρέπει να ενημερωθεί ο καταναλωτής και θα πρέπει να γίνει αυτό με συγχρηματοδότηση. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρόταση και ίσως εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε την κατανομή των πόρων μεταξύ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και αυτής που προέρχεται από εθνικές πηγές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να προωθούμε τις προτάσεις που πολύ σωστά εξέθεσε ο κ. Σταραμπέλα. Θα πρέπει να τελειώσουμε. Οι διερμηνείς μας έδωσαν λίγο παραπάνω χρόνο. Κύριε Ροσφόρ, ένα τελικό συνοπτικό σχόλιο. Ναι, ναι, ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι εδώ, που πήραν το λόγο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι τις 8 Μαΐου. 14 Μαΐου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες 29-30 Μαΐου. Οι συμβιβαστικές ελπίζω στις 19 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στις 20 Ιουνίου στην Επιτροπή. Έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η προθεσμία της τροπολογίας που δώσατε ίσως δεν είναι σωστή. Ε, είμαστε 6 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε πιο σύντομα. Α, συγγνώμη. 8 Μαΐου είναι πολύ πίσω. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες. Πιστεύω ότι και εσείς και οι σχεδοσυγητές περιμένετε κάποια απάντηση από την Επιτροπή, η οποία θα σας την υποβάλει. Ναι, 30 Μαρτίου βλέπω εδώ, είναι η σωστή ημερομηνία. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι 28 και 29 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες με φορτωμένο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ ή που μας παρακολουθήσατε.